το θέμα της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ειδικέ εκθέσεις σαν ένα χρήσιμο για τον νομοθέτη μέσο. Στόχος αυτής της ακρόασης είναι να μάθουμε από τις εμπειρίες των διεθνών ομολόγων μας και των κρατών μελών προσπαθώντας να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις των ελεγκτικών αυτών διαδικασιών. Να ακούσουμε τις απόψεις του Ευρωπαϊκού, του Αμερικανικού μάλλον αντίστοιχου ελεγκτικού συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μέσων δελικά που είναι διαθέσιμα για τη σωστή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων. Τέσσερις εμπειρογνώμονες θα δώσουν την άποψή τους για το θέμα αυτό. Στην πρώτη φάση της ακρόασης ο κύριος Κρίστοφερ Μιμ, Γενικός Διευθυντής για στρατηγικά θέματα, για θέματα στρατηγικής μάλλον, του Υπουργείου Εσωτερικών Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του GAO, θα μας μιλήσει για, τις, για τους ελέγχους σε επίπεδο επιδόσεων ε, της ομοσπονδιακής δαπάνης στις Ηνωμένε Πολιτείες, οι εμπειρίες του GAO και ο Ζω Μαρί Μπερτρό, γενικός εισηγητής και πρόεδρος του επιμελητηρίου των Γάλλων Ορκωτών Ελεγκτών, θα παρουσιάσει την δική του άποψη από πλευράς του δικού του επιμελητηρίου. Στο δεύτερο τμήμα ο Βίκτορ Καλντέιρα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, ε, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πάρει τον λόγο για τις διαφορετικές μορφές των ελέγχων και ο Αλγκύρντας Σέμετα, επίτροπος υπεύθυνος για τα τελωνία, τη φορολογία, τις στατιστικές και την καταπολέμηση της απάτης, θα μας μιλήσει για την χρήση των δίκτων σχετικά με τις επιπτώσεις έτσι όπως προσμετρούνται από την προοπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ακολουθήσει και μια γενική συζήτηση. Θα υπάρξει και η παρέμβαση του εισηγητή φυσικά ο κύριος Κυλακάκης, του κυρίου Σκυλακάκη. Θα ήθελα ξεκινώντας να δώσω το λόγο αμέσως στον συνάδελφό μου από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, τον κύριο George Lyon, ο οποίος θα μας μιλήσει για την προϋπτική ε, του προϋπολογισμού από ε, φυσικά την πλευρά της δικής του Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο για την εισαγωγή που έκανε. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ σαν εκπρόσωπος της Επιτροπής Προϋπολογισμών Είμαστε σαν υπεύθυνοι της Επιτροπής για την αδειοδότηση αν θέλετε των δαπανών, την έγκριση των δαπανών, εν είμαστε οι διατάκτες και επίσης προσπαθούμε να δούμε αν οι δαπάνες τις οποίες εγκρίνουμε είναι αποτελεσματικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και ποια είναι τα προγράμματα γενικότερα ε, στα οποία οι δαπάνε οι κοινοτικές οι ευρωπαϊκές επηρεάζουν θετικά. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα και για τις συζητήσεις ανάμεσα στις διαφορές ανάμεσα στους ελέγχους επί τη βάση της δραστηριότητας και στους ελέγχους επί τη βάση της επίδοσης, της αξιολόγησης της επίδοσης. Προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο και ποια μορφή ελέγχου είναι η καλύτερη για την αποτελεσματική χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Α, απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, υπάρχουν κίνδυνοι ε, τους οποίους έχει εντοπίσει το ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με την εισαγωγή ε, των αξιολογήσεων επί τη βάση της ε, καταμέτρησης της αποτελεσματικότητας της χρήσης των κριτηρίων. Και περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσω αυτά τα οποία θα μας πούν οι ομιλητές. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένω επίσης και την παρέμβαση ε, του εκπροσώπου της Αμερικανικής κυβέρνησης. Συναντηθήκαμε με το GAO όταν επισκεφθήκαμε τη Washington τον Ιούλιο και θα θέλαμε να μάθουμε ε, τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις με τον προϋπολογισμό τρία χρόνια μετά από την τελική αδυναμία, δεδηλωμένη αδυναμία του να καταλήξουν σε μια πλήρη συμφωνία για τα θέματα του προϋπολογισμού για πρώτη φορά στις Ηνωμένε Πολιτείε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμπροεδρεύσω εδώ και θα αναφέρω τις συζητήσεις σας στους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουμε όπως είπα τον κύριο Σκυλακάκη μαζί μας. Ο κύριος Σκυλακάκης είπα είναι εισηγητής για τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Well, uh, thank you. Σας ευχαριστώ. Βρίσκω ότι είναι σημαντική η σημερινή ακρόαση. Διότι επίκειται και οι ευρωπαϊκές εκλογές που θα είναι κέρια σημασίας γιατί γίνονται σε ένα κλίμα ευρωσκεπτικισμού σε όλη την Ευρώπη και στον Βορρά διότι ο κόσμος εκεί πιστεύει ότι τα χρήματά του δεν δαπανώνται σωστά και στον Νότο ή αλλού για άλλους λόγους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα, τα κονδύλια που δαπανώνται, δαπανώνται σωστά. Αυτό δεν είναι εύκολο. Εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, στα τελευταία χρόνια όπου έχω τη σχετική εμπειρία, διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και πολύ καλύτερα. Μπορούμε να δαπανίσουμε τα κονδύλια πολύ καλύτερα. Τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά τα διαχειρίζονται οι χώρες μέλη. Αυτό βέβαια δεν είναι δικαιολογία. Όταν εξετάσαμε την πρώτη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αυτό το αντιληφθήκαμε πολύ συγκεκριμένα. Για να δαπανηθούν τα χρήματα πιο αποτελεσματικά χρειάζεται και καλύτερο σχεδιασμός, λήψη καλύτερων αποφάσεων, αλλά και πολύ καλύτερος έλεγχος στο τέλος. Η έλεγχη αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας δεν είναι τυπική όπως είναι ορισμένη η έλεγχη της νομιμότητας και στις χώρες μας όπου έχουμε έλεγχο νομιμότητας ε, των δαπανών και ορισμένες φορές και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πάει και έχουμε δει σειρμούς μεγάλης ταχύτητας να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα αλλά μισοάδιοι και μάλιστα παράλληλα με αυτοκινητοδρόμους που είναι εντελώς άδειοι. Έχουμε πάει και έχουμε δει λιμάνια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μια πενταετία και ακόμα δεν έχουν συνδεθεί με τα σιδηροδρομικά δίκτυα ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν. τα ίσως είναι προφανή. Έχουμε επίσης προπετάσματα ε, για να μην περνάει ο θόρυβος των αυτοκινητοδρόμων δίπλα σε χωράφια, έτσι ώστε να μην οχλούν οι ίσως. Βλέπουμε λοιπόν πόσο άσχημα δαπανώνται ορισμένα από τα κονδύλια της Ένωσης και πρέπει να τροποποιηθεί. Την εμπειρία τη σχετική για το πώς μπορεί να γίνει αυτό δεν την διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότερες από τις χώρες μέλη μας αρκούνται σε ελέγχους νομιμότητας των δαπανών. Είναι λοιπόν σημαντικό να μπορέσουμε να βελτιώσουμε, να συλλέξουμε δηλαδή περισσότερη εμπειρία και να μπορέσουμε να δώσουμε ένα συνεχτικό μήνυμα στους Ευρωπαίους φορολογούμενους και ψηφοφόρους ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και αυτό να τους κάνει να έχουν πάλι μια πιο θετική άποψη για την Ευρώπη. Στην παρούσα ακρόαση, ή παρούσα ακρόαση καλύτερα, θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε και να υποβάλουμε τις ειδικέ εκθέσεις και επειδή εγώ έχω αναλάβει την εισήγηση για ορισμένες εξ αυτών, είναι πολύ καλοφτιαγμένες και πολύ χρήσιμες. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Θεόδωρε. Ας ακούσουμε τώρα τις εμπειρίες των Αμερικανών. Τον Κρίστοφερ Μιμ, Διευθυντή Στρατηγικών Θεμάτων στην ε, Υπηρεσία Οικονομικών της, ε, των ΗΠΑ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, μέλη της Επιτροπής. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα για να συζητήσω τις εμπειρίες μας στην Υπηρεσία Λογοδοσίας ε, του Δημοσίου, των ΙΠΑ. Όπως ξέρετε η αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε το έργο του Κογκρέσου, να ανταποκριθεί συνταγματικές του αρμοδιότητες και να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η απόδοση και η λογοδοσία του Ομοσπονδιακού κράτους προς όφελος του Αμερικανικού λαού. Οπότε συμφωνώ πλήρως με το σχόλιο του εισηγητού πως η χρηστή διοίκηση δεν είναι μόνο κάτι το τελετουργικό, είναι ουσιαστικό, είναι το πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνει τη σωστή προσοχή. Μετά την, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το Κογκρέσο ήθελε να έχει έλεγχο για τις ε, δαπάνες του Δημοσίου και το 1921 συνέστησε την υπηρεσία μας για να ελέγχει τις ομοσπονδιακές δαπάνες. Μετά τον ε, ε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεφύγαμε από τον ε, έλεγχο των τιμολογίων και κοιτάξαμε την απόδοση της ε, οικονομίας και των προγραμμάτων του κράτους. Οπότε ε, στη δεκαετία του 1960 αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο οι προσδοκίες από εμάς και ξεκινήσαμε να ελέγχουμε την απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Η νομοθεσία δε που πέρασε ε, ε, επέκτηνε ακόμη περισσότερο την νομοθετική βάση του έργου μας. Αυτό για εμάς ήταν μια μεγάλη αλλαγή στην δουλειά μας από αποκλειστικούς ελέγχους συμμόρφωσης προχωρήσαμε σε ε, αξιολόγηση της απόδοσης ε, των επενδύσεών μας. Εν ολίγης, από το να ρωτάμε το εάν πήγαν εκεί όπου όφυλαν τα λεφτά, ρωτούσαμε και το τι διαφορά έκαναν αυτές οι δαπάνες στη ζωή των πολιτών. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες λένε πως θα πρέπει να, έχουμε να παρέχουμε αντικειμενική ανάλυση έτσι ώστε το Κογκρέσο να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να κρίνει σωστά, να μειώσει το κόστος, να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και να συνεισφέρει στην λογοδοσία. Αυτός δε ορισμός συμμορφώνεται και με διεθνείς ε, προδιαγραφές ε, ελέγχου αποδοτικότητας επίσης. Εδώ πέρα εξυπονοείται πως ο ελεγκτής ξεκινά με ένα δημόσιο πρόγραμμα και από εκεί πέρα προχωρά. Κοιτάει δηλαδή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει αυτό το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής στη δουλειά μας βασίζεται σε κάποιες νομοθετικές εντολές, αιτήματα του Κογκρέσου και βεβαίως τις εντολές του Διευθυντού μας. Η εντολή μας λοιπόν βρίσκεται είτε σε νομοθεσία είτε σε εκθέσεις του Κογκρέσου που συνοδεύουν τους νόμους και επίσης όπως είπα έχουμε και συγκεκριμένα αιτήματα από το Κογκρέσο. Αυτές οι δύο κατηγορίες θα έλεγα πως αποτελούν γύρω στο 90% της δουλειάς μας. Δηλαδή είτε άμεσο αίτημα από τον νόμο είτε το Κογκρέσο μας ζητάει να ελέγξουμε κάτι. Επίσης εργαζόμαστε για όλε τι μόνιμε επιτροπές και 70% των υποεπιτροπών του Κογκρέσου. Το 2012, το οικονομικό έτος 2012, λάβαμε 924 ε, αιτήματα για έλεγχο και η συντριπτική πλειοψηφία από αυτό ήταν έλεγχο αποτελεσματικότητα. Το 2008 είχαμε μία διεθνή αναθεώρηση από ομοτήμους μας και επεσήμαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά που διέκριναν τη δική μας υπηρεσία από άλλες, ε, σε άλλες χώρες. Σε σύγκριση λοιπόν με τους ομολόγους μας κάνουμε μεγάλο αριθμό ελέγχων αποδοτικότητας, η πλειοψηφία των οποίων όπως σας είπα δεν είναι δική μας πρωτοβουλία αλλά τη δάει το Κογκρέσο. Επίσης σημειώθηκε πως απαντώντας στα αιτήματα του Κογκρέσου αποφασίζουμε εμείς το εύρος, τη μεθοδολογία, το χρόνο, τη στελέχωση και τη μέθοδο της δουλειάς μας. Δηλαδή μας ζητάει κάτι το Κογκρέσο αλλά δρούμε ανεξάρτητα. Επιπλέον έχουμε θετήσει κάποιες πρακτικές για να συμβιβάσουμε την δυνατότητα να αντιδρούμε σε αυτά τα οποία ζητάει το Κογκρέσο χωρίς να είμαστε κομματικοποιημένοι. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού όπου ε, το Κογκρέσο και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι ορίζουν τους βασικούς τομείς που πρέπει να διαχειρίζεται σωστά η, το δημόσιο. Ε, δηλαδή, η διαδικασία ξεκινάει και τελειώνει με το Κογκρέσο. Δηλαδή, ε, μας δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις και βεβαίως ε, κρίνουν και το έργο μας. Συναντιόμαστε με τα μέλη του Κογκρέσου και το προσωπικό τους ε, και βεβαίως ασχολούμαστε με τα ζητήματα που είναι δική τους προτεραιότητα. Δεύτερο, δεύτερη πρακτική είναι πώς εστιαζόμαστε κυρίως στους κινδύνους που υπάρχουν σε σχέση με κάθε αίτημα και επίσης σε τυχόν κινδύνους ως προς την ανεξαρτησία και το πώς θα το διαχειριστούμε και μπορούμε να πούμε πως έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Κάθε χρόνο παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις μας σε εκθέσεις και καταθέσεις ενώπιον του Κογκρέσου. Παραδείγματος χάρη το οικονομικό έτος 2012 είχαμε 650 εκθέσεις και καταθέσαμε επίση εκατοντάδες φορές στις διάφορες επιτροπές επιπλέον Κάθε μία από τις εκθέσεις μας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας ε, gao.gov δημοσιεύονται κάθε μέρα. Επίσης το οικονομικό όφελος από την δουλειά μας, το οποίο επαληθεύσαμε, ήταν 55,8 δισεκατομμύρια ε, δολάρια, δηλαδή 105 ε, δολάρια απόδοση για κάθε δολάριο που πάει στον προπολογισμό μας. Και βεβαίως έτσι ενισχύουμε και την λειτουργία του δημοσίου. Επίσης αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δίνουμε συνέχεια στις συστάσεις μας. Βλέπουμε πως γύρω στο 80% των συστάσεών μας εφαρμόζονται. Σαφώς ε, οι εθνικές ελεγκτικές υπηρεσίες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να δίνουν ε, στους ε, αξιωματούχους την ανάλυση που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Όμως τα προβλήματά μας σήμερα είναι παγκόσμια και απαιτούν διεθνή συνεργασία και διεθνείς λύσεις. Οπότε συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας ε, και τα ελεγκτικά συνέδρια, εθνικές υπηρεσίε από όλο τον κόσμο σε πάρα πολλά θέματα, όπως κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια οικονομική κρίση. Οπότε θα έλεγα πως οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσει ανά τον κόσμο γίνονται όλο και πιο πολύπλοκοι και διεθνείς. Είναι δηλαδή ζητήματα που δεν γνωρίζουν γεωγραφικά όρια, ούτε επίπεδα κυβέρνησης, ούτε ε, διαχωρισμούς κλάδων. Και βεβαίω οι δημοσιοπρεσίες βασίζονται σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και το μη κυβερνητικό τομέα και πρέπει να έχουν και τη διακριτική ευχέρεια Οπότε η γραμμή μεταξύ του κρατικού και μη κρατικού τομέα ε, καθίσταται όλο και πιο ισχνή. Επίσης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσμα τοπικών και παγκόσμιων προκλήσεων, αλλά και ζητήματα όπως ε, η προστασία της ασφάλειας των πολιτών, η φορολογική νομοθεσία, το ρυθμιστικό πλαίσιο, η δημόσια ασφάλεια π.χ. στον τομέα καταναλωτικών αγαθών, ιατρικών προϊόντων. Ουσιαστικά οποιοδήποτε σημαντικό αποτέλεσμα για το κοινό καλό απαιτεί διασυνοριακή και διυπηρεσιακή συνεργασία. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Προετοιμαζόμενοι για την πολυπλοκότητα» όρισε τέσσερις άξονες που θα είναι σημαντικοί τα επόμενα χρόνια. Ένας πολυπολικός κόσμος, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαμόρφωση πολιτικής από πολλοί ε, φορείς και η τεχνολογία. Προφανώς είναι γνωστές αυτές οι τάσεις και όπως ξέρετε η έκθεση κατέληξε ο νέος πολυπολικός κόσμος, το πολυεπίπεδο της διακυβέρνησης, οι πάρα πολλοί φορείς που διαμορφώνουν την νομοθεσία θα δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άμεσα ή έμεσα και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος κατακαιρματισμού της οικονομικής διοίκησης του ρυθμιστικού πλαισίου και υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η συνοχή, να υπάρχουν συστημικές αλληλεπικαλύψεις και συγκρούσεις. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή αξιολόγηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και οι ΙΠΑ. Η αξιολόγηση λοιπόν της αποτελεσματικότητας έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να δώσει αυτούς τους αλόγους αποφάσεις και στους πολίτες τις πληροφορίες και την ανάλυση που χρειάζονται για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον διασυνδεδεμένο κόσμο. Και φτάνουμε εδώ πέρα στο σημαντικότερο σημείο και το τελευταίο που θα ήθελα να πω. Για να συνεισφέρουμε στην διακυβέρνηση και στην διοίκηση του 21ου αιώνα θεωρούμε πως οι ελεγκτές θα πρέπει να εστιαστούν πολύ περισσότερο στην διοίκηση, στην διακυβέρνηση, δηλαδή να δουν τις διασυνδέσεις μεταξύ οργανισμών επιπέδων του κράτους, διαφόρων τομέων και μέσων πολιτικής. Αυτό είναι άρα ο λόγος για τον οποίο η αξιολόγηση αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας θα παραμείνει σημαντικό εργαλείο για εμάς και βλέπουμε πως θα πρέπει να αυξηθεί η έμφαση που δίνουμε σε αυτούς τους ελέγχους. Δηλαδή αντί να ξεκινήσουμε με ένα πρόγραμμα και να επεκτηνόμαστε σε ζητήματα συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, πρέπει να έχουμε ελέγχους που ξεκινάνε από το αποτέλεσμα και πάνε προς τα πίσω θα έλεγα. Δηλαδή να δούμε το ποιες είναι οι προσπάθειες που συνεισφέρουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις είναι η διαφορά του να κοιτάμε παραδείγματο, χάρη ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων και να δούμε πόσοι άνθρωποι ε, εκπαιδεύτηκαν και το να κοιτάμε την ανεργία και να δούμε το ποια είναι τα διάφορα προγράμματα που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα και πώς μεταξύ τους ε, διαπλέκονται. Και βεβαίως ε, και οι δύο αυτές προσεγγίσεις είναι χρήσιμες. Στην πράξη αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες για τη δουλειά μας που αναφέρονται στη γραπτή μου δήλωση που νομίζω σας έχει μοιραστεί. Πολλές, βεβαίως, από, πολλές φορές το αντικείμενο της δουλειάς μας αφορούν μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή πρόγραμμα. Υπάρχουν τρεις πρωτοβουλίες που είναι το πρόγραμμα υψηλού κινδύνου, η ετήσια έκθεση για τις άλλη επικαλύψεις και η έκθεση σύμφωνα ε, η έκθεση που οφείλουμε να κάνουμε σύμφωνα με την νομοθεσία του 2010 περί εξυγχρονισμού της διοίκησης μας δίνουν μια προοπτική για το πώς προσπαθούμε να αντιδράσουμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Να αναφερθώ λίγο σε αυτά, γιατί νομίζω πως είναι ενδεικτικά του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ πέρα αυτούς τους λαμβάνους αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα υψηλού κινδύνου. Τι κάνουμε, καταγράφουμε τις προκλήσεις διαχείρισης σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον διοίκησης. Ξεκίνησε το πρόγραμμα το 1990 και αρχικά στόχο είχε να εστιαστεί στις λειτουργίες εκείνης ε, της διοίκησης που είχαν ε, την μεγαλύτερη δυνατότητα για σπατάλη, απάτη και κακοδιοίκηση. Βεβαίως βλέπουμε συχνά πως ε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα κακών σχέσεων εργασίας με τρίτους όπως παραδείγματο χάρη αναδόχους έργων και ξεκινήσαμε έναν αναγκαίο μετασχηματισμό της διοίκησης. Σήμερα θα λέγαμε πως πάνω από τα δύο τρίτα των ε, τομέων εκείνων που είχαμε επισημάνει ως υψηλού κινδύνου που ήταν πάνω από χίλιοι είναι διατομεακοί. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ορίσαμε πως θα πρέπει να προστατευτεί περισσότερο το κράτος από την έκθεση σε κινδύνους κλιματικής ε, αλλαγής γιατί δεν βρίσκεται σε καλή θέση ως προς αυτό αυτή τη στιγμή το κρατσοβέως. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε υπηρεσία έχει την δική της αρμοδιότητα και δεν είναι η κλιματική αλλαγή εντός του χαρτοφυλακίου της, αλλά βρήκαμε πως θα μπορούσε να υπάρχει μια ενιαία συνεκτική στρατηγική και στο ομοσπονδιακό και στο πολιτιακό επίπεδο. Δεύτερον, αλληλεπικάλυψη, διπλή δουλειά και κατακαιρματισμός. Έχουμε εκδώσει τρεις ετήσιες εκθέσεις με αυτό το αντικείμενο που δίνουν μια συνολική εικόνα για πάνω από 162 τομείς και όρισαν 380 δράσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν και το Κογκρέσο και η διοίκηση για να μειωθεί, όπως είπα, ο κατακαιρματισμός και η αλληλεπικάλυψη, πέραν βεβαίως από τη μείωση του κόστους. Συνολικά οι τρεις αυτές εκθέσεις καλύπτουν κάθε μεγάλη ομοσπονδιακή υπηρεσία. Γεωργία, άμυνα, οικονομική ανάπτυξη, εκπαίδευση, ενέργεια κτλ. Και επίσης στην ιστοσελίδα μας ανεβάσαμε αυτό το οποίο λέμε τον μετρητή των δράσεων ε, για να δούμε ακριβώς που υπάρχουν οι συγκεκριμένες βελτιώσεις. Συνολικά το Κογκρέσο έχει σημειώσει κάποια πρόοδο. Το Μάρτιο φέτος ε, είπαμε πως γύρω στο 12% των σημείων που επισημάναμε είχαν αντιμετωπιστεί, 66% αντιμετωπιστεί εν μέρη και στο 21% δεν είχε υπάρξει κάποια αντίδραση. Υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες για την αξιολόγηση των επιδόσεων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Σαν παράδειγμα ε, υπάρχουν κάποιοι στόχοι υψηλής προτεραιότητας ε, οι οποίοι έχουν διασταυρούμενη προέλευση σε τομείς όπως η αηφορία, η προώθηση των εξαγωγών κτλ. Απαιτείται επίσης από τις μεμονωμένες υπηρεσίες να θέτουν τους δικούς τους στόχους και πέραν από τις δικές μας προσπάθειες να συνεισφέρουν στη βελτίωση της λειτουργίας τους. Όλα αυτά συνολικά θα βελτιώσουν την ομοσπονδιακή επίδοση. Η GAO επίσης περιοδικά θα παρουσιάζει περιληπτικά τις προσπάθειές της. Κυκλοφόρησε μια τέτοια έκθεση τον μήνα Ιούνιο και εκεί περιλαμβάνονται πάρα πολλά θέματα βέβαια τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και κυρίως η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Στις τελευταίες ε, τέσσερις δεκαετίες οι εμπειρίες μας στην ενσωμάτωση του performance audit στις ε, συνολικές μας μορφές λειτουργίας μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε την περιπλοκότητα των δημοσιονομικών είδαμε ότι οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν αλλαγές και στον δικό μας τρόπο ελέγχου ε, που αφορά ακριβώς την αξιολόγηση των επιδόσεων γιατί τα θέματα παρουσιάζονται πλέον με κατεπήγοντα χαρακτήρα. Όλα αυτά συζητιούνται και στο Κογκρέσο, συζητιούνται και σε επίπεδο πολιτικό αλλά και σε επίπεδο τεχνοκρατικό και εφόσον συμπεριλαμβάνεται και η άποψη των ορκωτών λογιστών γενικά και των ελεγκτών γενικότερα θα μπορέσουμε ίσως να βοηθήσουμε στην επίτευξη λύσεων. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Μίμα. Τώρα θα περάσουμε στη γαλλική εμπειρία μετά την αμερικανική. Θα δώσω το λόγο στο Ζω Μπερτρό, ο οποίος είναι γενικός εισηγητής του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρο που προσκαλέσατε το Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο να παρουσιάσει τις θέσεις του στα πλαίσια των ελέγχων της επίδοσης στο πλαίσιο ακριβώς της ακροάσεως την οποία οργανώνεται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Χαίρομαι που μιλάω μετά τον εκπρόσωπο του GAO με την οποία έχουμε πολύ στενές φιλικές σχέσεις και συμμετέχουμε και στον Διεθνή Οργανισμό Ελεγκτικών Συνεδρίων. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Διντιέ Μιγκό, μου ζήτησε να σας ζητήσω με τη σειρά μου συγγνώμη, δεν μπόρεσε να είναι παρόν γιατί συμμετέχει στην ακρόαση ε, στην, ε, της που οργανώνει η Επιτροπή η Αρμόδια της, της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Θα, ήταν, ε, θα ήθελε να είναι μαζί σας σήμερα, αλλά δυστυχώς θα προσπαθήσω να τον αντικαταστήσω όσο μπορώ καλύτερα. Πριν περάσω στην άποψη του συνεδρίου για το θέμα ακριβώς της αξιολόγησης των επιδόσεων θα ήθελα να σας μιλήσω για το τι συμβαίνει στη Γαλλία. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι, ανήκει σε επίπεδο διοικητικού δικαίου θα έλεγα ανεξάρτητο και από την εκτελεστική αλλά και την ομοθετική εξουσία. Προγραμματίζει ελεύθερα τις εργασίες της μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της 25ης Ιουλίου του 2001 και αυτό είναι και η εγγύηση της ανεξαρτησίας του. Το σύνολο των εργασιών του ελεγκτικού συνοδρίου ανταποκρίνονται στις τρεις μεγάλες αρχές της ανεξαρτησίας, της αντιπαράθεσης αλλά και ε, της συνέργειας. Οι δύο ιστορικές αποστολές του συνεδρίου είναι ο έλεγχος των, ε, των οικονομικών των, της δημόσιας διήγησης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που γίνονται από τους παρέδρους. Αυτό καλύπτει το σύνολο των δημοσιονομικών. Καλύπτει δηλαδή τις δαπάνες του κράτους και των υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτό, ε, των οργανισμών της δημόσιας ε, ε, γενικότερα και κοινωνικής προστασίας, ένας τεράστιος τομέας στη Γαλλία, πιο σημαντικός από το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, ε, και τους δημόσιους οργανισμούς και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Αν ο έλεγχος των λογαριασμών και της διαχείρισης των περιφερειακών οργανώσεων ασκείται όχι από μας, αλλά από αντίστοιχες ομόλογες περιφερειακές ομάδες, οι οποίες και αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, Παρ' όλα αυτά εμείς σαν κεντρικό ελεγκτικό συνέδριο σε στενή συνεργασία με αυτές τις περιφερειακές υπηρεσίες παρακολουθούμε το σύνολο των τοπικών ε, οικονομικών δραστηριοτήτων του Δημοσίου. Θα δημοσιεύσουμε σε ένα μήνα περίπου μια πρώτη συνθετική έκθεση για αυτό που ονομάζουμε ε, τοπικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών. Ταυτόχρονα εμείς ε, ε, ελέγχουμε και τον, την χρήση κάποιων ιδιωτικών κονδυλίων τα οποία λαμβάνονται από δημόσιους οργανισμούς ως δωρεές ε, μετά από εκκλήσεις προς την δημόσια γενεοδορία ή την γενεοδορία του κοινού, κάτι το οποίο βέβαια δίδει στους συγκεκριμένους πολίτες ε, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Η δραστηριότητα του ελεγκτικού συνεδρίου ασκείται σε δύο τομείς. Καταρχάς, ο έλεγχος συμβατότητας, μέσω του οποίου ε, το συνέδριο ελέγχει την κανονικότητα των δημοσιονομικών και λογιστικών ενεργειών και διασφαλίζει τον σωστό σεβασμό των πρακτικών διαχείρισης. Ε, μια διαδικασία δικαστική μπορεί να οδηγήσει ε, τον έλεγχο να θέσει σε αμφισβήτηση και την προσωπική ευθύνη ε, των ορκωτών λογιστών του δημοσίου, δηλαδή των παρέδρων. Σχετικά με τους τάκτες δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ή να θέσουμε σε κίνδυνο τη δική τους ευθύνη, αλλά μπορούμε να ζητήσουμε τη διαμεσολάβηση ε, του ε, τακτικού δικαστηρίου που ασχολείται με θέματα δημοσιονομικά. Ε, συμπροεδρεύεται από τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνοδρίου και αποφασίζει για τις κυρώσεις και για τα πρόστιμα στους διατάκτες που έχουν κηρυχθεί ένοχοι. Έτσι λοιπόν κάνουμε και τις λεγόμενες ελεγκτικές διαδικασίες ε, ε, αξιολόγησης των επιδόσεων. Ελέγχουμε δηλαδή τη σχέση ανάμεσα στα μέσα που εμπλέκονται και στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα μάλλον. Και τη σχέση ανάμεσα στα αποτελέσματα που έχουν ε, επιτευχθεί και στα αποτελέσματα τα οποία είχαν τεθεί σαν στόχος. Εδώ είναι η αποτελεσματικότητα. Θα επανέλθω σε αυτά. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ελέγχου θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το σύνολο των δημοσιονομικών για, ένα από τα τρία, για κάθε ένα από τα τρία υποσύνολα. Δηλαδή το κράτος, την κοινωνική ασφάλιση και τέλος τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Έχουν προσταθεί, προσθεθεί πρόσφατα και δύο άλλες αποστολές. Καταρχάς η πιστοποίηση ε, των λογιστικών του κράτους και του ε, γενικού καθεστώτος της κοινωνικής ασφάλισης μετά από το 2006 όπως επίσης και η αρρωγή προς το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση στα πλαίσια της αξιολόγησης των δημοσίων πολιτικών ε, που ξεκίνησε μετά από την συνταγματική αλλαγή του 2008 για την άσκηση αυτών των τεσσάρων αρμοδιοτήτων, τον έλεγχο, την κρίση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση χρησιμοποιούμε 411 άτομα ελεγκτές, από τους οποίους 230 δίκαστες και 211 άτομα τα οποία είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι εργασίες μας έχουν σαν στόχο να δώσουν εγγυήσει για το τακτό και την ποιότητα της δημόσιας διαχείρισης. Επιτρέπουν επίσης να διαφωτιστούν οι πολιτικοί σε σχέση με τις ανεπάρκειες πιθανώς της δημόσιας διαχείρισης και να ξεκινήσουν με προτάσεις μεταρρύθμισης. Γι' αυτό συνοδεύουμε συστηματικά τις παρατηρήσεις μας με συστάσεις ε, για τις οποίες ελέγχουμε εφόσον έχουν εφαρμοστεί μετά από λίγα χρόνια. Η ετήσια έκθεση ε, του ε, ελεγκτικού συνοδρίου είναι μια παρουσίαση θα έλεγα και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις μας τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση των αποστολών του Ελεγκτικού συνεδρίου θα ήθελα να επανέλθω στη σημαντική μεταρρύθμιση των γαλλικών δημοσιονομικών στοιχείων εδώ και 12 χρόνια. Μια μεταρρύθμιση που επιτρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια των δημοσίων λογαριασμών, μια πιο καθαρή και λειτουργική παρουσίαση της δημοσιονομικής κατάστασης και της περιουσιακής κατάστασης του γαλλικού κράτους και μια ενίσχυση των εξουσιών των ελεγκτικών του Κοινοβουλίου. Η μεταρρύθμιση αυτή τροποποίησε κατά πολύ τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ε, θα έλεγα η αποστολή του ελεγκτικού συνεδρίου. Για πάνω από 40 χρόνια τα γαλλικά δημοσιονομικά μετά τον πόλεμο δηλαδή τον δεύτερο καθορίζονταν από το διάταγμα της Δευτέρας Ιανουαρίου του 1959. Ήταν ο οργανικός νόμος των δημοσίων δαπανών οι δαπάνες αυτές παρουσιαζόντουσαν ανακεφάλαιο και αναυπουργείο ανάλογα με την οργάνωση του συγκεκριμένου Υπουργείου χωρίς να υπάρχουν όλες οι δυνατότητες συζήτηση των στόχων της δημόσιας δαπάνης. Η αποτελεσματικότητα δηλαδή της δημοσίας δαπάνης δεν ήταν υπολογίσιμη. Ο νέος οργανικός νόμος, ο οποίος έγινε δεκτός την 1η Αυγούστου του 2001, ο λεγόμενος Λόλφ, νόμος Λόλφ, Τότε ο πρόεδρος μας Μιγκό ήταν γενικός εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών ε, της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, οδήγησε στις απαιτούμενες καινοτομίες του δημοσιονομικού και λογιστικού γαλλικού πλαισίου. Από το 2006 και μετά ο προϋπολογισμός του κράτους οργανώνεται σε αποστολές και σε προγράμματα. Μία αποστολή διυπουργική ή απλά υπουργική περιλαμβάνει ένα σύνολο προγραμμάτων που συγκλίνουν σε μια συγκεκριμένη δημόσια πολιτική. Ένα πρόγραμμα ομαδοποιεί τις πιστώσεις που έχουν σαν, στέχη, σαν στόχο συγγνώμη, την κινητοποίηση μιας δράσης σε ένα συγκεκριμένο Υπουργείο. Οι πιστώσεις αυτές δικαιολογούνται μέχρι το τελευταίο ευρώ και φυσικά όλα αυτά ε, σε ένα όριο αναυπουργείο. Η παρουσίαση αυτή του προϋπολογισμού διαφωτίζει το Κοινοβούλιο για την τεκμηρίωση των προτινομένων δαπανών, για τους στόχους των δαπανών αυτών και ενημερώνεται το Κοινοβούλιο και για τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Στα πλαίσια αυτού του νόμου η επίδοση μιας δημόσιας πολιτικής υπολογίζεται από τους στόχους, τους αντικειμενικούς στόχους, τους επιμέρους στόχους σε επίπεδο τριών κατηγοριών. Αποτελεσματικότητα κοινωνικο-οικονομική, για τον πολίτη, ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στο χρήστη και αποδοτικότητα, δηλαδή βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μέσων. Προσμετράται επίσης από συγκεκριμένους αριθμητικούς δείκτες. Κάθε στόχος συνοδεύεται από ένα δείκτη και γίνεται αντικείμενο παρουσίασης στα πλαίσια μιας ετήσιας παρουσίασης των επιδόσεων για κάθε ένα από τα προγράμματα και συνδέεται φυσικά με τον κρατικό προϋπολογισμό σε ετήσια βάση ε, άλλωστε γίνεται και ένας έλεγχος κάθε τμήματος του προϋπολογισμού ε, είναι οι λεγόμενες αιτήσει εκθέσεις. Ο νόμος ΛΟΛΦ έχει σαν στόχο την υπευθυνοποίηση των διαχειριστών του δημόσιου χρήματος. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος καθορίζουν ε, τους στόχους τους και προσμετρούν τα αποτελέσματά τους. Μπορεί να ζητήσουν την τροποποίηση της κατανομής των ποσοστών των κονδυλίων που έχουν στη διάθεσή τους, ε, χωρίς βέβαια αυτό να θίξει άλλες κατηγορίες δαπανών λειτουργικών, δηλαδή λειτουργίας, επέμβασης και επένδυσης. Ο νόμος Λόλφ έχει τρεις βασικούς στόχους. Καταρχάς τον καλύτερο καθορισμό των δημοσιονομικών πολιτικών την καλύτερη προσπάθεια καθορισμού της στρατηγικής τους και τα πλαίσια τους. Επιβεβαιώνει την ευθύνη αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα περιθώρια δράσης τους και δίδοντάς τους νέα μέσα διαχείρισης. Και τέλος βελτιώνουν τα αποτελέσματα της δημόσιας δαπάνης και σε επίπεδο αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας προς τον πολίτη ακριβώς μέσω της καλύτερης διατύπωσης των στόχων που κατατίθενται στο Κοινοβούλιο και της εισαγωγής των δικτών επίδοσης που επιτρέπουν την προσμέτρηση των αποτελεσμάτων. Ο νόμος Λόλφ επέβαλε στο κράτος να λαμβάνει υπόψη ε, την ανάγκη διατήρησης μάλλον όχι μόνο μια συγκεκριμένης λογιστικής των εσόδων και των δαπανών αλλά και μιας γενικής λογιστικής μεθόδου του συνόλου αυτών των δράσεων για να υπάρχει πάντα η πλήρης εικόνα της οικονομικής κατάστασης του κράτους. Ο νόμος Λόλφ ε, εμπιστεύθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο τον έλεγχο του τακτού, της ειλικρίνειας και της πιστότητας των δημοσίων λογαριασμών. Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύθηκε από την ενίσχυση των δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου που του επιτρέπουν να ασκήσει καλύτερα με τη συνεργασία του ελεγκτικού συνεδρίου τις εξουσίες του στον τομέα του ελέγχου και της αξιολόγησης. Ο νόμος Λόλφα από το 2001 και μετά και ο οργανικός νόμος της Δευτέρας Αυγούστου 2000 2005 που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση της κοινωνικής δαπάνης που είναι όπως είπα τεράστια δαπάνη, μεγαλύτερη από τον υπολογισμό λειτουργίας του κράτους. Ε, ενισχύουν οι νόμοι αυτοί λοιπόν τις αρμοδιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου και συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου που είναι η αρρωγή στο κοινοβούλιο και, τον, και την κυβέρνηση. Ε, ο νόμος Λόλφ και η συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση Λόλφ ΛΟΛΦ-ΕΣ που αφορά τις κοινωνικές δαπάνες περιλαμβάνει έξι ετήσιες εκθέσεις που στηρίζουν τις ενέργειες της κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, δύο εκθέσεις πιστοποίησης των δημοσίων λογαριασμών και του καθεστώτος που αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Η πιστοποίηση αυτή έχει σαν στόχο το να δοθεί μια συγκεκριμένη έλογη εγγύηση της ποιότητας των λογαριασμών και κατά συνέπεια της εικόνας που δίδουν για την οικονομική κατάσταση του κράτους, της περιουσίας του κράτους, των χρεών του κράτους και των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται. Πέραν από, αυτούς, από αυτές τις εκθέσεις πιστοποίησης έχουμε και τρεις εκτελεστικές εκθέσεις. Μία ετήσια έκθεση για τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους γενικά. Συνοδεύεται από αναλύσεις της εκτέλεσης του προϋπολογισμού αναποστολή και αναπρόγραμμα. Παρουσιάζεται πριν από τις 30 Μαΐου σε ετήσια βάση. Παρουσιάζουμε 60 περίπου αναλυτικές εκθέσεις, ε, τεκμηριώνοντας την έκθεση αυτή, για να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο για το τακτό της δημοσιονομικής εκτέλεσης, ε, ε, την αξιολόγηση των επιδόσεων, το υποστηρίξιμο ημί όλων των αποστολών του προϋπολογισμού του κρατικού στη φάση ακριβώς εξέτασης από το Κοινοβούλιο του ετήσιου ε, των, λογαριασμών του προηγούμενου έτους. Παρουσιάζουμε επίσης ε, και ένα νόμο για την χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Η έκθεση αυτή παρουσιάζεται πριν από την εξέταση από το Κοινοβούλιο του νόμου που αφορά τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης για το επόμενο έτος ασχολείται με τις επιδόσεις της κρατικής παρέμβασης στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της βιωσιμότητας των κοινωνικών δαπανών. Προστίθεται εδώ μια έκθεση η οποία αφορά τις δανειοδοτήσεις από τον ε, προϋπολογισμό όταν το, όταν το κράτος είναι υπεύθυνο να πάρει πιστώσεις ανάμεσα σε δύο περιόδους δημοσιονομικές. Τέλος παρουσιάζουμε μια έκθεση το μήνα Ιούνιο για την κατάσταση και τις προοπτικές των δημοσιονομικών, του συνόλου των δημοσιονομικών. Η έκθεση αυτή βασίζεται κυρίως, ε, βασίζει μάλλον την συζήτηση προσανατολιστική η οποία γίνεται στο Κοινοβούλιο στις αρχές του καλοκαιριού για τον επόμενο προϋπολογισμό. Η επόμενη έκθεση για τις τοπικές αρχές και περιφερειακές αρχές θα συμπληρώσει τις ετήσιες εκθέσεις για τα δημοσιονομικά της Γαλλικής Δημοκρατίας έτσι ώστε και οι τρεις τομείς ε, της δημόσιας διοίκησης να καλυφθούν πλήρως. Πέραν αυτών των ετησίων εκθέσεων οι Επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου δηλαδή της Εθνικής Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, ζητά συγκεκριμένες έρευνες από το ελεγκτικό συνέδριο και έχουμε στη διάθεσή μας εμείς 8 με 12 μήνες για να τις παραδώσουμε. Το 2012 ε, δόθηκαν 15 τέτοιες εκθέσεις έρευνες σε ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές για διάφορα θέματα όπως το Εθνικό Κέντρο Κινηματογραφίας, η συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου ε, το κόστος της επανένταξης της γαλλικής δημοκρατίας στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ κτλ. Ο καθορισμός των θεμάτων αυτών των ερευνών είναι αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο ελεγκτικό συνέδριο για να μην θυγεί ε, ο ελεύθερος προγραμματισμός των εργασιών μας. Αυτή τη στιγμή δοθούν στο Κοινοβούλιο οι εκθέσεις αυτές, οδηγούν σε μια ακρόαση από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, των ε, μελών του ελεγκτικού συνεδρίου, τη παρουσία εκπροσώπων των δημοσίων υπηρεσιών με τους οποίους ασχολείται η έκθεση. Και όλα αυτά δημοσιεύονται. Η συνταγματική μεταρρύθμιση της 23 η Ιουλίου του 2008 έχει επιβεβαιώσει και ενισχύσει το ρόλο του δικαστηρίου εισάγοντας ένα νέο άρθρο το 47.2 στο γαλλικό σύνταγμα. Λέγει το άρθρο 47.2. Το ελεγκτικό συνέδριο συνδράμει το κοινοβούλιο στον έλεγχο της δράσης της κυβέρνησης ταυτόχρονα συνδράμει το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση στον έλεγχο της εκτέλεσης των δημοσιονομικών της χώρας και στην εφαρμογή ε, της χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης όπως και στον τομέα της αξιολόγησης των δημοσίων πολιτικών. Μέσω αυτών των δημοσίων εκθέσεων το ελεγκτικό συνέδριο συμμετέχει και στην σωστή ενημέρωση των πολιτών. Το ελεγκτικό συνέδριο το γαλλικό λοιπόν έχει ε, μια μεγάλη αρμοδιότητα. Βοηθά το κοινοβούλιο, βοηθά ε, την κυβέρνηση και ενημερώνει σωστά και τους πολίτες. Ταυτόχρονα συνεισφέρει και στην αξιολόγηση των αναγκών των δημοσίων πολιτικών. Πώς τώρα προχωρά στην επίτευξη αυτών των ελέγχων επιδόσεων. Αν δείτε τις τέσσερις αποστολές τις οποίες ασκεί το Συμβούλιο, δηλαδή έλεγχος, κρίση, επιβεβαίωση και αξιολόγηση, ε, ιδιαίτερα ο έλεγχος και η αξιολόγηση συνδέονται άμεσα με τον έλεγχο επιδόσεων. Αν και βέβαια και η δικαστική πλευρά και η επιβεβαιωτική είναι απαραίτητες. Ο όρος ε, audit de performance, έλεγχος των επιδόσεων, δεν χρησιμοποιείται στο γαλλικό δίκαιο παραδοσιακά και μιλάμε για έλεγχο της σωστής χρήσης των δημοσιονομικών. Όταν ε, το συνέδριο αποφάσισε να προχωρήσει στον έλεγχο ενός δημοσίου οργανισμού σαν παράδειγμα, οι ερευνητές ε, του Δικαστικού ε, Συμβουλίου εξετάζουν σε βάθος την κατάσταση των λογαριασμών του οργανισμού, τις διάφορες κατηγορίες δαπανών, λειτουργία, επενδύσεις κτλ. Ο έλεγχος δεν σταματά στην εξέταση της διαχείρισης στρίκτο σένσο. Ε, αφορά επίσης και την δημόσια πολιτική ευρύκαιρα στην οποία συνεισφέρει ή εφαρμόζει ο υποέλεγχο οργανισμός. Εμείς σαν συνέδριο δεν καθορίζουμε τους στόχους και τους δείκτες, αλλά αναφερόμεθα στους στόχους και στους δείκτες τους οποίους έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση ε, μέσω του προϋπολογισμού ή που καθορίζονται με συμβατικό τρόπο ανάμεσα στο κράτος και τον δημόσιο οργανισμό στα πλαίσια μιας σύμβασης στόχων και μέσων, όπως λέγεται, ε, για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της δημόσιας παρέμβασης. Μπορεί να αποφασίσει ε, το συνεδρίο ότι οι δείκτες αυτοί δεν είναι οι σωστοί ε, σε σχέση με τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί και να προτείνει διαφορετικούς. Η έλεγχη του, Συμβουλίου, του ελεγκτικού συνεδρίου συγγνώμη, ε, οδηγούν σε προσωρινές ε, συστάσεις και μετά από μια αντιπαράθεση και διαβούλευση δημοσιεύονται οι τελικές συστάσεις. Ταυτόχρονα προχωρούμε και στην αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών και με δική μας πρωτοβουλία και με πρωτοβουλία ε, των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι αξιολογήσεις αυτές αφορούν μια συγκεκριμένη πολιτική δημόσια στο σύνολό της και όχι σε μια επιμέρους πολιτική ρύθμιση ή σε μια οργάνωση. Οι συγκεκριμένες αυτές αξιολογήσεις ελέγχουν τους στόχους που επιδιώκονται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται και έχουν σαν στόχο την εγκυρότητα της εφαρμογής μιας δημόσιας πολιτικής σε επίπεδο συνεκτικότητας, αποδοτικότητας και χρησιμότητας. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των αξιολογήσεων αυτών δείχνουν ότι το συνέδριο χρησιμοποιεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, χρησιμοποιεί αναλυτικά μέσα ιδιαίτερα αναλυτικά, όπως ακριβώς τα δειγματολόγια, και συμμετέχει γενικά στην εξέταση της εφαρμογής της πολιτικής αυτής και προσπαθεί να αποκαταστήσει τους δεσμούς που μπορεί να εξηγήσουν τα καλά ή τα λιγότερο καλά αποτελέσματα τα επιδιωχόμενα αυτής της πολιτικής. Είναι εγκάρσια αυτή η διάσταση, αυτή η αντιμετώπιση, είναι εταιρική, είναι συγκριτική και δράζεται στην έρευνα συγκεκριμένων μεθόδων προόδου. Διαφορετικά από τον έλεγχο των επιδόσεων, η αξιολόγηση επιλέγει και οικοδομεί τους δείκτες οι οποίοι θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι. Συμπληρώνει την ικανότητα του ελεγκτικού συνεδρίου να αξιολογήσει την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών. Πρόκειται όμως για προσπάθειες οι οποίες είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και γι' αυτό είναι και λίγες. Κάνουμε 4 ή 5 γενικότερες εξηγολογήσεις κατέτος. Ε, το συνέδριο προχώρησε το 12 σε μια αξιολόγηση της πολιτικής κατά της χρήσης των προϊόντων καπνού, όπως επίσης και της πολιτικής στήριξης δημιουργίας επιχειρήσεων. Οι αξιολογήσεις αυτές παραγγέλθηκαν ε, στην Επιτροπή Αξιολόγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Προχωρήσαμε εμείς και ε, στον έλεγχο της πολιτικής βοήθειας στα βιοκαύσιμα, όπως επίσης και των ασφαλιών ζωής. Συμπερασματικά, σε σχέση με τις ετήσιες εκθέσεις της LOLF και της LOLF-SS, κοινωνική ασφάλιση, που ήδη προανέφερα, θα καταλήξουμε στις εξής παρατηρήσεις. Καταρχάς, παρατηρήσεις α, τελικές, οι οποίες απευθύνονται άμεσα στον ελεγχόμενο οργανισμό, που δεν δημοσιοποιούνται αλλά μπορεί αν θέλει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να τις μάθει. Μετά, γενικότερες αναφορές οι οποίες καταντίθενται στην κυβέρνηση και στις δημόσιες υπηρεσίες και οι οποίες συστηματικά μεταδίδονται στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση και δημοσιεύονται σε μία προθεσμία δίμηνη με την απάντηση του συγκεκριμένου Υπουργού κατέτος. Στέλνουμε στην κυβέρνηση περίπου 30-40 τέτοιου είδους συνολικές αποφάσεις οι οποίες δημοσιοποιούνται οι περισσότερες τουλάχιστον. Η ίδια διαδικασία για εκθέσεις οι οποίες αφορούν τους δημόσιους οργανισμούς, τις δημόσιες επιχειρήσεις, όπως επίσης ε, ενημερώνονται η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο και εδώ. Έχουμε και μια ετήσια δημόσια έκθεση και τις λεγόμενες θεματολογικές δημόσιες εκθέσεις, 15 ε, περίπου που αφορούν συγκεκριμένα θέματα και καλύπτουν έναν τομέα συγκεκριμένο. 15 περίπου το χρόνο. Απευθύνονται στις δημόσιες αρχές αλλά γενικότερα στους πολίτες και καλύπτουν έναν τομέα ευρύτερο ε, δημιουργώντας μια σύνθεση σαν παράδειγμα όλων των ελεκτικών δραστηριοτήτων μας. Τους τελευταίους 6 μήνες έχουμε δημοσιεύσει εκθέσεις στους εξής τομείς. Αγορά εργασίας, εδαφική οργάνωση, διαχείριση του ε, εκπαιδευτικού δυναμικού, δημόσιες πολιτικές υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διάσωση της τράπεζας, δέξια κτλ. Το ελεγκτικό συνέδριο ασκεί στη Γαλλία λοιπόν συγκεκριμένες ευρύτατες αρμοδιότητες λόγω της ενίσχυσής της εδώ και 15 χρόνια. Η υιοθέτηση του νόμου ΛΟΛΦ το 2001 επέτρεψε την τροποποίηση σε βάθος της παρουσίασης του προϋπολογισμού από το κράτος, δίδοντας συγκεκριμένους δείκτες για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας δαπάνης. Όπως και αν και όπως το είπε το συνέδριο το 2011, Δέκα χρόνια μετά τον ΛΟΛΦ η προοπτική μιας νέας διαχείρισης των μεγάλων δημοσίων πολιτικών με μεγαλύτερη ευθύνη και με έλεγχο των αποτελεσμάτων έχουν επιβραδυνθεί από κάποιες ε, διστακτικές αντιλήψεις στην ε, κυβέρνηση ε, αν και βέβαια ο ρόλος, ο καθοριστικός ασκείται από το Κοινοβούλιο και πρέπει να ασκηθεί ακόμα πιο αυστηρά. Με τους πολλαπλούς ελέγχους της ε, η υπηρεσία μας έχει μπορέσει να βοηθήσει τις ε, δημόσιες πολιτικές. Πέρα από τις παρατηρήσεις και συστάσεις που στέλνουμε στις δημόσιες αρχές, βασικός μας στόχος είναι να ξέρει ο πολίτης πώς χρησιμοποιείται το δημόσιο χρήμα, όπως το προβλέπει το άρθρο 15 ε, της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολίτη, σύμφωνα με το οποίο η κοινωνία έχει δικαίωμα να ζητήσει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται από τη δημόσια διοίκηση το δημόσιο χρήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. κύριε Jean-Marie και τώρα έχετε ώρα να θέσουμε ερωτήσεις να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην συζήτηση εφόσον το επιθυμείτε. Πρώτο έχω εγγεγραμμένο τον εισηγητή κ. Σκυλακάκη. Και θα ακολουθήσει ο κύριος Μπαλτσίτης, η κυρία Γιάρα Σέντερ, και μετά από αυτήν ο κύριος Μίλτερ. Άρα πρώτος εσείς κύριε Σκυλακάκη. Θα ήθελα να θέσω πρώτα μια ερώτηση στον κύριο Μιμ για το πρόγραμμα υψηλού κινδύνου, High Risk Program. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που εξήγησατε. Έχω προσπαθήσει την τελευταία διετία να εισαγάγω στη δική μας υπηρεσία πολέμης απατών, Όλαφ, να τους εισαγάγω λοιπόν την έννοια ότι πρέπει από μόνοι τους με δική τους πρωτοβουλία να ερευνούν σε τομείς υψηλού κινδύνου, χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω λίγο περισσότερο για, τα, όσα κάνετε. Δεύτερο, όταν έχετε εντοπίσει τους high risk areas, το επόμενο σας βήμα ποιο είναι. Απάντηση, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Το πρόγραμμα υψηλού κινδύνου άρχισε μέσα από μια απογοήτευση που αισθανόταν το Αμερικανικό Κογκρέσο ότι δηλαδή είχαν ε, σημειωθεί ένας αριθμός σκανδάλων υψηλής ορατότητας και επίσης ε, προβλήματα και στους ίδιους τους οργανισμούς μειωμένης αποδοτικότητας και αναρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι το High Risk Program σχεδιάστηκε να πάρει είναι μόνο 30 αυτή τη στιγμή που έχουν ε, τα, τα όργανα που έχουν αυτά και να τους δώσει την ορατότητα που χρειάζονται έτσι ώστε να, μπορούν, να μπορέσουν να αρχίσουν να ασχολούνται μαζί τους όπως είπα ενημερώνεται και το Κογκρέσο για την εποπτεία και πέραν της ζωής κάθε κοινοβουλευτικής θητείας όταν εμείς εντοπίζουμε κάτι ως υψηλού κινδύνου αρχίζει βέβαια έλεγχος πριν να εντοπιστεί ο τομέας αυτός. Έτσι οι ελεγκτές εγκύπτουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό. Και εμείς εργαζόμαστε ανεξάρτητα μένα, αλλά πολύ στενά με άλλους αξιωματούχους, καθώς και με αξιωματούχους του Κογκρέσου, για να καθορίσουμε συγκεκριμένα ποιες ενέργειες πρέπει να αναλυφθούν για να αντιμετωπιστεί η ρίζα των προβλημάτων. Για παράδειγμα, στη συνεργασία με τρίτους όπως εργολάβους ή υπεργολάβους σε πολύ περίπλοκες, για παράδειγμα, προημήθειες οπλικών συστημάτων κλπ. Έτσι παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά για να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν. Υποβάλλουμε αναδιετία έκθεση είναι περίπου 30 οι τομείς όπως είπα υψηλού κινδύνου, αλλά κάθε ένας από αυτούς έχει εν τέλει στην έκθεση 3-4 σελίδες. Αλλά το βασικό είναι να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Είτε εμείς είτε το Κογκρέσο. Τι πρέπει να κάνει στα πλαίσια του νομοθετικού του έργου για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έρχονται από αυτού του τομεί κινδύνου. Προβλήματα τα οποία καμιά φορά εκκρεμούν από πολύ καιρό, άλλα επανέρχονται κάθε τόσο και εξακολουθούμε και ασχολούμαστε με αυτά. Μπορέσαμε την τελευταία φορά να βγάλουμε από τον κατάλογο αυτό κάποιου τομεί, προσθέσαμε άλλου, αλλά πάντως έχουμε εξυπηρετήσει στη διάρκεια του προγράμματο αυτού πολύ καλά την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Προεδρεύων. Σα ευχαριστώ και εσείς κύριε Μπαλτσίτης τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ νόμιζα ότι θα μιλήσει πρώτος ο πρόεδρος Καλντέρα πριν, από, πριν να μπορέσω να θέσω εγώ την ερώτηση. Πάντως και εγώ θέλω να ρωτήσω τον Αμερικανό εκπρόσωπο. Έχετε περιπτώσεις όπως εξή. εξής. Εσείς καλείστε να εκτελέσετε ένα συγκεκριμένο καθήκον. Δεν μπορείτε όμως να υποβάλλετε τα συμπεράσματά σας στο Κογκρέσο, γιατί κάποια πολιτεία δεν μπορεί να σας δώσει τα απαραίτητα δεδομένα. Δεύτερο, κατανόησα καλά ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του οργάνου σας συνδέεται ή αν έρχεται περίπου στο ποσό των 550 εκατομμυρίων ε, δολαρίων και είπατε ότι ένα δολάριο ε, αποδίδει 105. Πώς λειτουργεί ε, ο οργανισμός σας. Ζητείτε συγκεκριμένους δείκτες και ποιοι είναι οι στόχοι για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση απάντηση. Σας ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση για τα δεδομένα. Βέβαια είναι από τις πιο θεμελιώδεις προκλήσεις για τους ελέγχους μας και πολύ συχνά ε, καταναλώνει πολύ χρόνο. Συχνά μάλιστα δεν είναι μονάχα θέμα με τις, ε, των πολιτιών μας δηλαδή να μας παράσχουν τα απαραίτητα ε, στοιχεία και άλλοι οργανισμοί έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι οι οργανισμοί είτε κολυσιεργούν είτε αρνούνται να μας παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Το θέμα είναι περισσότερο και είμαι βέβαιος ότι και οι εδώ παρόντες συνάδελφοι μου θα αντιμετωπίζουν ενδεχομένω το πρόβλημα αυτό, ότι οι οργανισμοί έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες καλής αποδοτικότητας, κόστους κλπ. Και πολύ συχνά οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις για να μπορέσουν να μας πούν ποιο ακριβώς είναι το κόστος ενός προγράμματος που έχουν αναλάβει. Εμείς έχουμε κάποιες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά και την αξιοπιστία των δεδομένων που λαμβάνουμε και οποιασδήποτε πληροφορίες λαμβάνουμε από άλλους οργανισμούς και αποδοτικότητας του κόστους. Αυτά μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο και να μην διαθέτουμε επαρκή χρόνο εμείς τότε βέβαια αυτό το θέτουμε υπόψη του Κογκρέσου. Πολλές από τις συστάσεις μας έχουν την έννοια αυτή. Λέμε στους οργανισμούς ότι χρειάζεστε καλύτερα, πιο στέρεα πληροφοριακά στοιχεία, όχι μόνο για τους ελεγκτές. Θέλω να ρωτήσω τον program manager, να μπορώ να τον ρωτήσω δηλαδή, αν δεν γνωρίζεις, αν δεν έχεις καλές, στέρεες πληροφορίες για το κόστος, πώς θα μπορείς να διαχειριστεί το πρόγραμμα. Είναι λοιπόν βασική ευθύνη αυτή. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το έτοιμά μας για τον προϋπολογισμό. Εμείς περνούμε από την ετήσια ενιάυσια, δηλαδή έγκριση των δαπανών μας, του προϋπολογισμού μας δηλαδή από το Κογκρέσο, αλλά απευθείας από αυτό. Ο Υπουργός της κάθε φορά υποβάλλει τον προϋπολογισμό μας για τα όργανα μας και συνεργαζόμενοι μαζί του εξετάζουμε και πολλές λεπτομέρειες. Πόσα χρήματα τον πήρατε από τον CEO την προηγούμενη, τι απόδοση είχατε κτλ. Τι κάνετε για να εξορθολογήσετε τις επιχειρήσεις σας, όπως και όλοι οι άλλοι οργανισμοί στις ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν και σε όλο τον κόσμο μεγάλη πίεση να εξορθολογήσουν τις υπηρεσίες τους, να δίνουμε έγκαιρα πληροφορίες σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και εμείς να δίνουμε έγκαιρα και στην μορφή που χρειάζονται οι νομοθέτες τις προφορίες που απαιτούνται. Διεξάγουμε τη συζήτηση αυτή. Είμαστε τυχεροί επειδή το έργο μας είναι επιτυχές. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές μας. Αλλά είμαστε και σε ανταγωνισμό με άλλους που ε, τραβούν χρήματα από τον προϋπολογισμό. Έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό βέβαια και έχω βάλει και στην δήλωσή μου ένα σχετικό φύλλο. Έχουμε και performance report που λέει πώς ανταποκριθήκαμε στους στόχους μας και για την Επιτροπή Προϋπολογισμών αλλά και για τις επιτροπές που μας εποπτεύουν. Ευχαριστώ, λέει ο Προεδρεύων. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για τις δύο παρεμβάσεις που έγινα και ίσως να θέσω κάποια ερωτηματικά στον εκπρόσωπο του GAO. Τι εμπειρίες έχετε από τη διαχείριση των μηχανισμών που έχουν σχέση και με τα δημοσιονομικά αλλά και με την οικονομική κρίση. Ε, ενώ τι έγινε όταν εθνικοποιήθηκαν ορισμένα πιστοτικά ίδρυματα. Είναι κάτι το οποίο συμμετέχει στον εξάντε έλεγχο των δημοσιονομικών τα χρήματα που δόθηκαν δηλαδή στις τράπεζες αυτές ή μόνο εκ των υστέρων ενημερωθήκατε και κάνατε τον έλεγχο της χρήσης των συγκεκριμένων πιστώσεων. Δεύτερον, ο οργανισμός αυτός είναι δημόσιος και ασχολείται μόνο με το δημόσιο προϋπολογισμό ή έχει την δυνατότητα να ελέγχει και ιδιωτικές πιστώσεις και ιδιωτικά ταμεία όπως ακριβώς μπορεί σε κάποιες, με κάποιες προϋποθέσεις να κάνει ε, ο Γάλλος ομόλογός σας. Τώρα, ε, ασχολείστε και ε, συμμετέχετε στις εργασίες όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών ανάλογα με τη θεματολογία ή καλείστε μόνο να ενημερώνετε την Ολομέλεια. Και έχετε επίσης πρόβλημα με τον έλεγχο των προγραμμάτων όπου υπάρχει ε, θέμα στο οποίο συμμετέχουν στη χρηματοδότησή του όχι μόνο ο προπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, ομοσπονδιακός, αλλά και χρήματα από άλλους οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, σαν παράδειγμα. Και τέλος, η κατάρτιση των παρέδρων. Τι ακριβώς κάνετε. Ε, έχετε κάποιο πρόγραμμα διαβίου κατάρτισης ε, των ελεγκτών σας, των παρέδρων σας. Δεν ξέρω, μπορώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις και στον κύριο Μπερτρόν. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά πάντα με την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, με ποιο τρόπο το Γαλλικό Ελεκτικό Συνέδριο ελέγχει τον γαλλικό προϋπολογισμό ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σωτηρίας των Τραπεζών. Γνωρίζετε ότι πρόκειται για έναν οργανισμό λουξεμβουργιανού δικαίου. Ε, πώς οργανώσατε εσείς τον έλεγχο αυτών των δημοσίων κονδυλίων ε, στα πλαίσια ενός μηχανισμού που είναι διακυβερνητικός και άλλου τύπου. Ε, ταυτόχρονα εσείς είστε ξεκάθαρα ένας δημόσιος οργανισμός, ελέγχετε τα δημόσια οικονομικά, είπατε όμως ότι μερικές φορές καλείστε ε, να χρησιμοποιείτε και εξωτερικούς ελεγκτές. Αυτό είναι κάτι το, ε, που αυξάνεται στη χρήση των εξωτερικών ελεγκτών. Με ποιο τρόπο δημιουργείται αυτή τη σχέση, τίθεται αυτή η σχέση. Κανονικά ένα ελεγκτικό συνέδριο κανονικά ε, ελέγχει εκ των υστέρων, αλλά το γαλλικό ε, ελεγκτικό συνέδριο επί τη βάση του νόμου Λόλφ, ε, όπως μας είπατε από το 2001, μπορεί και εκ των προτέρων να συμμετέχει στον προγραμματισμό των δαπανών της κυβέρνησης. Είπατε εσείς ότι η ελευθερία προγραμματισμού είναι εγγύηση για την ελευθερία λειτουργία σας, αλλά ταυτόχρονα Αυτά στα οποία αναφερθήκατε έχουν σχέση γενικά με την προστασία των συμφερόντων των Γάλλων πολιτών. Ο... Δεν ασχολείστε με τον έλεγχο θεμάτων που δεν ενδιαφέρουν την γαλλική κοινωνία. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν με ποιο τρόπο εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στην καθημερινή συζήτηση η οποία γίνεται για τα δημοσιονομικά. Και τέλος, μας δώσατε τα θέματα με τα οποία ασχολείστε και μέσω ακριβώς της εμπειρίας ε, του ελεγκτικού σας συνεδρίου ε, πώς επικοινωνείτε με το κοινό. Ε, έχετε δυνατότητα να επηρεάσετε μόνο μέσω της απλής ενημέρωσης, μέσω της ενημέρωσης ανακατηγορίες, της εκπαίδευσης, με ποιο τρόπο μπορεί το κοινό να συμμετέχει μαζί σας. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω ε, ε, είπατε ότι είναι διαφανής ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε. Μας δώσατε κάποιες εξηγήσει και βλέπω και εγώ τον κύριο Καλδέιρα ο οποίος πολλές φορές είναι θύμα κάποιων προβλημάτων στον τομέα αυτό. Ε, εσείς χρησιμοποιήσατε στα πλαίσια της εξέτασης συγκεκριμένων προγραμμάτων συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να είναι αναγνώσιμα από το κοινό, εννοεί η ομιλήτρια. Και πώς, εν πάση περιπτώσει, προετοιμάζετε τελικά σε επίπεδο πρακτικό τις εκθέσεις σας. Ευχαριστώ, κυρία μου. Όπως είδατε, αλλάξαμε προεδρία εδώ, αλλά τελείως δημοκρατικά και γαλήνια θα παρακαλέσω, μιας και ακούστηκαν ερωτήσεις και προς τον κύριο Μιμ και τον κύριο Μπερτράν, παρακαλέσω πρώτα τον κύριο Μιμ να απαντήσει και μετά ας απαντήσει ο κύριος Μπερτράν αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Αν ε, σε κάτι δεν σας απαντήσω, ελπίζω να απαντήσω όλα, δεν το κάνω από πρόθεση να με ξαναρωτήσετε. Το πρώτο, για τους ελέγχους για την οικονομική κρίση. Παίξαμε κέριο ρόλο ενημερώνοντας το Κογκρέσο για δύο πτυχές. Πρώτα την νομοθεσία διαχείρισης, το Trouble Asset Relief Program δηλαδή, TARP, ανά δίμηνο υποβάλαμε εκθέσεις στο ε, κοινοβούλιο μας, πώς χρησιμοποιούνταν τα κονδύλια κλπ. Δεύτερο, για το πρόγραμμα κινήτρων τάξος 860 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Φλεβάρι του 2009. Πάλι εκεί ένα δίμηνο εξετάζαμε πώς χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά οι πολιτείες. Και κάθε 45 ημέρες, στο τέλος κάθε τριμήνου, μιλούσαμε για τις προβλέψεις ε, στην απασχόληση, για τον αριθμό θέσεων απασχόλησης δηλαδή που δημιουργούνταν. Άρα είχαμε τρεις ξεχωριστές απαιτήσεις ελέγχων. Όσον αφορά τώρα ε, να προωθήσουμε την μεγάλη ε, νομοθεσία μετά από αυτό το ΤΑΡΠ που σας είπα, έχουμε 40 ξεχωριστές νομοθετικές απαιτήσεις για να υποβάλουμε εκθέσεις για το πώς διαμορφωνόταν η νομοθεσία, αν ήταν έγκαιρη, εάν είχε το ποθούμενο αποτέλεσμα το φάσμα δηλαδή. Η μεγάλη διαφορά με τον συνήθι τρόπο λειτουργίας του GAO είναι ότι μας αναγκάζουν να εργαζόμεθα σε ρυθμό διμήνων. Ήταν πολύ δύσκολο, ωστόσο ήταν υγιές από μια άποψη, με την έννοια ότι επέτρεψε στο Κογκρέσο να λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο περίπου. Ρωτήσατε επίσης για εκ των προτέρων ε, εν αντιθέσει με το εκ των υστέρων διεξαγωγή ελέγχων. Συχνά μέλη του Κογκρέσου μας ζητούν να σχολιάσουμε νομοθεσία, ιδίως για νέα προγράμματα, αν είναι καλά σχεδιασμένα κλπ. Από ό,τι καταλαβαίνω σχετικά με το τι γίνεται εδώ, αυτά που κάνουμε δεν είναι τόσο πειθαρχημένα και τυποποιημένα. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας βουλευτής σε εμά που σκέφτεται να υποβάλει κάποιο σχέδιο νόμου και να μας πει για πες μου GAO βασισμένος στο μέχρι τώρα έργο σου πού μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει η πρόταση. Μας ενδιαφέρει περισσότερο εάν η εν λόγω σχεδιαζόμενη νομοθεσία εμπεριέχει και κάποια εντολή προς εμάς για τη διεξαγωγή ελέγχων. Αυτό μας ενδιαφέρει και τότε ερχόμαστε σε επαφή με το προσωπικό του γερουσιαστή ή του βουλευτή για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κάνουμε λοιπόν λίγο και το εξάντε, αλλά περισσότερο σε βάση ad hoc και ανεπίσημη. Τώρα, για τους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς έχουμε αρμοδιότητα και, και ευθύνη να ακολουθούμε τη δημόσια δαπάνη όπου και να πάει. Το ομοσπονδιακό δολάριο δηλαδή ή την ομοσπονδιακή επιρροή. Αλλά δεν θα εξετάσουμε αποκλειστικά μόνο πώς δαπανώνται ιδιωτικά κονδύλια. Ένα ενδιαφέρον πράγμα ε, αυτά που σας είπα προηγουμένως, ΤΑΡΠ είναι τα κεφάλαια που εισέρευσαν και σε πρώην δημόσιους οργανισμούς και επομένως για μας παρέμειναν μέσα στο ε, πεδίο αρμοδιοτήτων μας. Εφόσον χρειάζεται να πάμε σε κάποιον βουλευτή και να πούμε εδώ μπορούμε να σας απαντήσουμε ή όχι, αν υπάρχει δηλαδή κάποια διασύνδεση με το ομοσπονδιακό επίπεδο. Για την ερώτησή σας, αν εργαζόμαστε για λογαριασμό όλων των επιτροπών ή μόνο για την Ολομέλεια. 70% των υποεπιτροπών και όλες οι επιτροπές του, του Κοινοβουλίου μας, 160 μαρτυρίες συνολικά, αυτές είναι από κυρίως τέσσερις επιτροπές. Το δικό μου χαρτοφυλάκιο λοιπόν σημαίνει ότι έρχομαι εγώ σε επαφή κυρίως με τους ομολόγους σας στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Αλλά οι συνάδελφοί μου θα πάνε να δούνε και αυτούς που ασχολούνται με το financial services, ενδεχομένως ε, απασχόλησης, ενδεχομένως άμυνας. Βάζουμε ας πούμε να ε, συνεργαστούν εμπειρογνώμονες με εμπειρογνώμονες σε τα ειδικά θέματα. Τώρα, για προβλήματα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι διεθνείς οργανισμούς Ακολουθούμε, όπως είπα, τις ομοσπονδια... τα ομοσπονδιακά κονδύλια όπου και να πάνε. Εκεί που γίνεται πιο περίπλοκα τα πράγματα, για παράδειγμα προγράμματα βοήθειας για αναπτυσσόμενες χώρες, τα αμερικανικά κονδύλια μπορεί να αποτελούν μόνο ένα τμήμα και ούτε καν καθοριστικό της συγκεκριμένη επένδυσης. Παρ' όλα αυτά και εκεί έχουμε την ευθύνη για να ελέγξουμε. Ίσως γνωρίζετε ότι το στρατηγείο των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το κτίριο ε, ανακαινίζεται και κάνουμε ελέγχους και σε αυτό. Και με άλλη μου ιδιότητα εκτός GAO είμαι επικεφαλής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που υποστηρίζει την Γενική Συνέλευση για ένα, θέμα, για ένα ε, αριθμό θεμάτων εποπτείας και αποδοτικότητας. Είναι λοιπόν και άλλος ένας τρόπος αυτός με τον οποίο εμπλέκεται το GAO. Όσον αφορά την εκπαίδευση, ναι, αυτό για μας παίζει σημαντικό ρόλο. Οι έλεγχοι μας απαιτούν να έχουμε τουλάχιστον 80 ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αναδιετία. Αυτό είναι και απέτηση και αν δεν φτάσω αυτές τις 80 ώρες θα πρέπει να βγω εκτός γραμμής, offline και θα πρέπει για να επανέλθω να συμπληρώσω τις, ε, την εκπαίδευσή μου. Κάνουμε μεγάλη ε, επένδυση για να πάνε οι άνθρωποι μας σε ειδικέ διαδέξεις, σεμινάρια κτλ. Είναι έρθουν ειδικοί να μας ε, ενημερώσουν γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους με υψηλά προσόντα. Τέλος, για διαφάνεια. Εμείς συνομιλούμε με οποιονδήποτε δημοσιογράφο ή μέλος του κοινού σχετικά με το συνεχιζόμενο έργο μας για το ποιοι είναι οι στόχοι της δουλειάς αυτής, ποιος ζήτησε την άσκηση του ελέγχου, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, και για το τι πρέπει να γίνει. Αν μας ρωτήσετε για κάτι λέμε ότι «Ε, το κάνουμε για λογαριασμό του τάδε βουλευτή ή μπορούμε να σας πούμε ότι θα το κάνουμε το τάδε πράγμα την άνοιξη του 2014. Και εάν εσείς ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, θα πούμε και γιατί γίνεται. Όταν έχει γίνει η δουλειά αυτή και όταν έχει υποβληθεί η έκθεση, μπορείτε να την κρατήσετε εμπιστευτική για 30 ημέρες. Μετά από αυτό, βγαίνει στην ιστοσελίδα και συνομιλούμε με οποιονδήποτε. Εμείς δεν κάνουμε συνεντεύξεις τύπου κλπ. Αλλά ευχαρίστως συνομιλούμε με το κοινό ή με τα μέσα σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων μας. Τέλος, όλα τα έγγραφα εργασίας μας κλπ. εκτός εάν είναι εμπιστευτικά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου Freedom of Information και θεωρούμε ότι άλλωστε αυτό είναι και η ορθή πρακτική. Είχαμε περιπτώσεις όπου πολίτες ή άλλοι ζήτησαν πρόσβαση στα έγγραφά μας και την χορηγήσαμε. Πιστεύουμε ως οργανισμός ότι χρειαζόμαστε διαφάνεια στην εκτελεστική εξουσία και ε, θεωρούμε ότι έχουμε πρωτοπόρο ρόλο. Σας ευχαριστώ κοιτώντας την κυρία Γιάλα Σέντερ νομίζω πως είναι πραγματικά ικανοποιημένη με την απάντησή σας. Ναι, χαμογελούσε. Λοιπόν, τώρα τον λόγο έχει ο κύριος ε, Μπέρτραν και βεβαίως είναι και ο κύριος Μέτα εδώ πέρα, ο Επίτροπος. δω αν μπορώ να είμαι το ίδιο αποτελεσματικός όπως ο Κρίστοφερ Πρώτα για τον έλεγχο του συνεδρίου, πώς παρεμβαίνει το συνέδριο, πώς παρεμβαίνει μάλλον για την οικονομική κρίση, με δύο τρόπους. Αφενός σφαιρικά, με τους ελέγχους που διεξάγουμε πολλές φορές τον χρόνο για το σύνολο των δημοσίων οικονομικών. Είπα ότι υποβάλλουμε έκθεση για την εκτέλεση του κρατικού προπολισμού τον Μάιο, τον Ιούνιο υποβάλλουμε έκθεση για το σύνολο των δημοσίων οικονομικών και επανερχόμεθα στην ετήσια έκθεσή μας πάλι για το σύνολο των δημοσίων οικονομικών τον μήνα ε, Φεβρουάριο κάθε χρόνο. Και με την ευκαιρία αυτή εγκύπτουμε σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά και βέβαια η οικονομική κρίση είχε άμεση επιπτώσει στον κρατικό προϋπολογισμό με τι πιστώσει που ανοίχθηκαν ή με τι εγγύσει που δόθηκαν από τον ίδιο προϋπολογισμό. Εκφραστήκαμε εκεί. Πρώτο, έλεγχη. Δεύτερο, έλεγχη τη τράπεζα τη Γαλλία, τη κεντρική δηλαδή γαλλική τράπεζα, η οποία συναπαρτίζει την Ευρωπαϊκή. Ε, την ελέγχουμε. Ελέγξαμε και το πακέτο βοήθειας στις γαλλικέ τράπεζε και ιδίω τις εγγύησεις που έχει δώσει το γαλλικό κράτος και έχουμε υποβάλει πλειό, πλήθος εκθέσεων σχετικά που έχουν δημοσιευτεί. Επίσης, η νέα συνθήκη του Μαρτίου του 2012 για την δημοσιονομική εποπτεία εμπλέκει και αμέσω και αμέσως το ελεγκτικό συνέδριο, αμέσως για την ανάλυση των δημοσιονομικών, όπου Μάιο και Ιούνιο αναφερόμαστε και στο πρόγραμμα σταθεροποίησης το οποίο έχει υποβληθεί και στα ευρωπαϊκά όργανα από τον Απρίβη και εξάλλου η Γαλλική Εθνοσυνέλευση έχει ιδρύσει και ένα όργανο το οποίο είναι το Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών και στηρίζεται στην εργασία και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το όργανο αυτό έχει ως αποστολή να τοποθετείται για τις οικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίζει την πολιτική της η γαλλική κυβέρνηση για, την, για το σχεδιασμό του προϋπολογισμού. Ήδη η γαλλική κυβέρνηση καταθέτει τις μεγάλες γραμμές του προϋπολογισμού του 2014, επ' αυτού εκφράζει άποψη για τα μακροοικονομικά. Εκεί ξεφεύγουμε από το καθαρό χώρο αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου γιατί κοιτάζουμε προς το μέλλον. Δεύτερο, τι κάνουμε με τους εμπειρογνώμονες. Προσφεύγουμε όλο και περισσότερο σε εμπειρογνώμονες και μάλιστα με δύο τρόπους. Αφενός για ιδιαίτερα θέματα όπου προσλαμβάνουμε εμπειρογνώμονες και ενδεχομένως τους αποζημιώνουμε, ε, μπαίνουν στις ε, ομάδες ελέγχων μας και επίσης διαβολευόμαστε με τους ε, εμπειρογνώμονες όλο και περισσότερο για θέματα που βλέπουμε. Η πρακτική συνίσταται στο να ερχόμαστε σε επαφή με τους εμπειρογνώμονες και να ε, οργανώνουμε συζητήσεις μαζί τους. Παρεμβαίνουμε εκ των προτέρων εξάντε, όχι. Το ελεγκτικό συνέδριο προβαίνει σε ελέγχους εκ των υστέρων. Άρα ε, αμέσως όχι. Ωστόσο, όπως και ο συνάδελφός μας της Αμερικανικής GAO, έχουμε σχέσεις με τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και όταν συζητούμε ένα θέμα, μετά για παράδειγμα από μια παραγγελία μιας ε, κοινοβουλευτικής επιτροπής, μας ζητείτε η γνώμη, μας ερωτούν σχετικά με το εφαρμόσιμο των λύσεων που ε, επιλέγει ε, η κυβέρνηση και αν μπορούν να επαληθευτούν υποθέσεις ενδεχομένως για την αποτελεσματικότητα ή την κανονικότητα. Κάθε έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου συνοδεύεται σήμερα και από κατάλογο συστάσεων. Τέταρτο, πώς επιλέγουμε, είναι ανεξάρτητο το συνέδριο. Εγώ τόνισα ότι η ανεξαρτησία αυτή σημαίνει και ελευθερία προγραμματισμού. Το συνέδριο δεν δημοσιεύει τον προγραμματισμό του. Τι κάνει. Ε, κινούμε από μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική η οποία επικυρωποιείται κάθε χρόνο και η οποία μας επιτρέπει να επιλέγουμε έναν αριθμό στρατηγικών προτεραιοτήτων για τους ελέγχους που θα ασκήσουμε τα επόμενα χρόνια για τα δημόσια οικονομικά. Μετά βασιζόμαστε σε αναλύσεις κινδύνου στους διαφόρους τομείς αναλύουμε αυτό το στρατηγικό ε, προβληματισμό σε τριετή σχέδια, τα οποία βεβαίως ενημερώνουμε κάθε έτος και στη βάση αυτή κάνουμε μετά έναν ετήσιο προγραμματισμό που εγκρίνεται στα τέλη του έτους, τον Δεκέμβριο δηλαδή του έτους και έχει ισχύ για το επόμενο έτος, ε, περιλαμβάνοντας σε αυτόν τον προγραμματισμό και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου που μας έρχονται συνήθως το φθινόπωρο. Συζητούμε δηλαδή τις παραγγελίες που λαμβάνουμε από τα κοινοβουλευτικά όργανα, συνήθως για 18 μήνες ή για 2 χρόνια γιατί τα θέματα των ερευνών βέβαια χρειάζονται συνήθως κάποιο χρόνο. Με ρωτήσατε ακόμη για τις συνολικές επισκοπήσεις. Το ελεγκτικό συνέδριο δημοσιεύει από τούδε πρόσφατη εξέλιξη αυτή και μετά από την συνταγματική αναθεώρηση του 2008 τα ουσιαστικά στοιχεία των εκθέσεών μας. Δημοσιεύουμε τι σημαίνει κυρίως την ιστοσελίδα. Αρχίζουμε απευθύνοντας τις εκθέσεις στους ελεγχόμενους οργανισμούς και σε ένα διάστημα μηνών στις αρμόδιες επιτροπές της Γαλλικής Έθνος Και ταυτόχρονα τα βάζουμε επιγραμμικά μαζί με ένα σύντομο ανακοινοθέν που εξηγεί το περιεχόμενο της παρεμβάσεως. Για τις θεματικές τώρα δημόσιες εκθέσεις, εκεί οργανώνουμε συνεντεύξεις τύπου και κάθε σχετική έκθεση συνοδεύεται από ένα ανακοινωθέν τύπου και από μια επισκόπηση 10-15 ε, σελίδων οι οποίες ε, εξηγούν σύντομα το θέμα και όπως είπα ε, ενημερώνεται ο τύπος. Τέλος με ρωτήσατε για την διαφάνεια. Κατανόησα ότι σας ανησυχεί η διαφάνεια ιδίως των ελέγχων. Έχουμε τρεις μεγάλες αρετές για παράδειγμα. Ε, ε, ε, διαφάνεια κλπ. Τώρα, συλλογικό, συλλογικός χαρακτήρας δεν είμαστε ιεραρχικό όργανο. Όλες οι εκθέσεις εγκρίνονται από ένα συλλογικό σώμα τουλάχιστον τριών παρέδρων. Και βεβαίως τίθεται υπόψη και του Προέδρου και ψηφίζονται. Επίσης, κατά μολία. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχει μία προσωρινή έκθεση, αυτή ε, ε, τίθεται υπόψη του ελεγχόμενου οργανισμού, ο οποίος καλείται να αντιδράσει και στη βάση αυτών των σχολείων του πλέον ε, εγκρίνει το συνέδριο την τελική έκθεση. Περιλαμβάνουμε πάντοτε τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων και ελεγχόμενων οργανισμών και στην ιστοσελίδα. Άρα, πρώτο τμήμα είναι η έκθεση και δεύτερο η απάντηση του Υπουργείου ή οποιοδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου που διαλαμβάνεται μέσα στην έκθεση. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο είμαστε απολύτως διαφανείς. Thank you very much, Mr. Bertrand. Σας ευχαριστώ. Ο Γιάνν Μιλτερ είναι ο επόμενος ομιλητής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια απλή ερώτηση έχω. Κάθε χρόνο έχουμε εδώ πέρα την ε, παρουσίαση του κυρίου Καλντέρα, του πρόεδρου του ελεκτικού συνεδρίου, για το πώς εφαρμόστηκε ο προϋπολογισμός. Ε, υπάρχει ένα ακρονίμιο, μια ε, διαβεβαίωση όπως λέγεται και η απάντηση είναι απλή αν το ελεγκτικό συνέδριο δίνει ναι ή όχι μια τέτοια σωστή διαβεβαίωση και 19 χρόνια σειρά η απάντηση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι αρνητική και βεβαίως ε, ο λόγος είναι πως ε, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιτρέπεται ένα ποσοστό λάθος 2% στον προπολογισμό. Το ερώτημά μου είναι πολύ απλό. Εάν υποθέσουμε πως Εφαρμόζομαι το όριο του 2% στον προπολογισμό των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα θα ήταν θετικό και το ίδιο ερώτημα για τη Γαλλία επίσης. Thank you very much because you are asking, Mr. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε νομίζω θα ήθελα να επεκταθεί, αν δεν σας πειράζει. Θα μιλήσω γερμανικά. Ένας συνεργάτης μου ερευνήσε και είπε πως έχετε ένα ποσοστό λάθους 10%. Ε, ε, ισχύει αυτό. Σας ευχαριστώ. Εάν ε, δεν σας πειράζει, θα ήθελα να προτείνω να αλλάξουμε λίγο τη μεθοδολογία μας γιατί ξέρω ότι ο κύριος Μιμ κάνει ό,τι μπορεί. Ε, απαντάει πολύ αναλυτικά. Οπότε ας ακούσουμε άλλη μία ερώτηση ε, από τον κύριο Αντιπρόεδρο και μετά να απαντήσει ο κύριος Μιμ. Proposing short, with was concerned mainly answers, not questions. Ε, ε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου προς τον ε, κύριο Μιμ. Όσον αφορά τις ομοσπονδιακές δαπάνες πρόνοια, υγεία και εκπαίδευση. Τα περισσότερα, τις περισσότερες δαπάνες τις κάνουν οι πολιτείες, όχι το ομοσπονδιακό κράτος. Το ερώτημα λοιπόν που έχω και αφορά και το ερώτημα ενός συναδελφού. Όταν κάνετε έλεγχο, φαντάζομαι πως έχετε εξουσίες να μπείτε όπου θέλετε και να ζητήσετε ε, πληροφορίες από τις ε, πολιτείες. Ε, μπορείτε μετά και να επιβάλλετε κυρώσεις, να διορθώσετε λάθη, να διασφαλίσετε κάπως τη σωστή λειτουργία και αν αρνηθούν γιατί κάποιες ε, πολιτείες αρνήθηκαν παραδείγματος χάρη να εφαρμόσουν το νέο νομοσχέδιο περί παροχής υγείας το Ομπάμα και το λεγόμενο παρά το ότι είναι ονδιακή νομοθεσία. Και εδώ πέρα έχουμε μια παρόμοια κατάσταση γιατί μεγάλο μέρος του ποσοστού του σφάλματος ε, είναι ζήτημα των κρατών μελών. Γιατί οι κυβερνήσεις εκτελούν τα... οι εθνικές κυβερνήσεις εκτελούν τα προγράμματα. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Βλέπω λοιπόν, δεν θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια ερώτηση. Ο κύριος Μιμ. Και μην ξεχνάτε πως θα έρθει και ο κύριος... Ε, θα ακούσουμε και τους κύριους Καλτέρα και σε μετά, έτσι, να έχουν και αυτοί λίγο χρόνο. Ναι, ναι, βεβαίω, για να είμαι σύντομο. Να ξεκινήσω από το τέλο. Δεν έχουμε δυνατότητα και αρμοδιότητα επιβολή, Έχουμε μόνο την πειθό μα και ενώπιον του Κογκρέσου και ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστούν οι συστάσεις αυτές αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι. Όσον αφορά το 10% ποστό λάθους αυτό το οποίο το ανάλογο στι Ηνωμένε Πολιτείε θα ήταν ε, κάποια χρεωστήτω καταβληθέντα θα λέγαμε ποσά. Υπάρχουν ε, ε, νομικές απαιτήσεις που ορίζουν ένα ποσοστό το οποίο είναι 2,5% για δαπάνες πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια ή από 100 εκατομμύρια δολάρια ξεκινώντας από το οικονομικό έτος 2014, δηλαδή τον Οκτώβριο. Και τον Οκτώβριο θα μειωθεί στο 1,5% το ποσοστό. Οπότε εξορισμού από την ομοθεσία οτιδήποτε πάνω από αυτό θεωρείται πως δεν συμμορφώνεται. Τη δουλειά δεν την κάνουμε εμείς, την κάνουν οι εσωτερικοί ελεγκτές της κάθε υπηρεσίας και οι γενικοί επιθεωρητές. Ικανοποιηθήκατε με αυτή την απάντηση και ο κύριος Χιλακάκης. Οπότε, ποιο είναι το μέσο ποσοστό σφάλματος για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ε, δεν το έχω, θα το στείλω στην Επιτροπή σας για τα πρακτικά, δεν το έχω πρόχειρο. Ε, η πρόκληση είναι πως υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα, οπότε το κοιτάμε ένα πρόγραμμα. Έχουμε, αδείγμα τους χάρη, ε, τα τέλη του Medicare προγράμματος παροχής υγείας έχει ένα 8,5% ε, ποσοστό ε, σφαλμάτων, γύρω στα 30 δισεκατομμύρια δηλαδή το χρόνο. Οπότε η στρατηγική που κάνουμε με τις υπηρεσίες βεβαίως και τους γενικούς επιθεωρητές τους πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακτήσουμε τα λεφτά αυτή τη στιγμή έχουν εκταμιευθεί δύσκολο και αναποτελεσματικό απλά πρέπει να υπάρξει περισσότερος ε, έλεγχος ε, και ε, κυρίως πριν εκταμιευτούν τα λεφτά εκεί πέρα δίνουμε βάρος τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ. Κατόπιν θα ακούσουμε τον ε, κύριο Καλντέρα και τον κύριο Επίτροπο. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας παρουσιάσετε εσείς ε, τα σχετικά. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, εσείς κύριε Σιγητά, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι και εσείς αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ που με επιτρέπετε να λάβω μέρος στην ακρόαση που φαίνεται να στρέφεται γύρω από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Άρα για μένα έχει μεγάλη σημασία να μπορέσει να απευθύνει το λόγο και το συνέδριο στην Επιτροπή σας. Μου ζήτησαν, ε, μου ζητήσατε να μιλήσω για ένα θέμα η διεξαγωγή ελέγχων για νομιμότητα και κανονικότητα από την σκοπιά του ελεγκτικού συνεδρίου. Θυμήθηκα λοιπόν ότι πρόσφατα ο καθηγητής Λέβη σε άλλη παρόμοια ακρόαση είχε υποβάλει το εξής ερώτημα. Ποιο είναι πιο σημαντικό, η αποδοτικότητα ή η κανονικότητα, η νομιμότητα δηλαδή. Αν συμφωνείτε θα έλεγα ότι μάλλον πρόκειται για μια ψευδοεπιλογή. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι το θέμα. Συμμόρφωση, νομιμότητα, απόδοση. Για το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να ισχύουν και τα δύο για έναν συγκεκριμένο αριθμό λόγων. Πρώτα υπάρχει ένας νομικός λόγος. Η συνθήκη λειτουργίας της Ένωσης λέει καθαρά ότι το συνέδριο ελέγχει εάν κάθε έσοδο έχει εισπραχθεί και κάθε δαπάνη έχει εκτελεστεί με νόμιμο και κανονικό τρόπο και αν η διαχείριση υπήρξε χρηστή. Αυτή είναι η εντολή μας. Και μετά ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει επίσης την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ως εφαρμογή των αρχών της ε, οικονομίας αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Επομένως, η εντολή του ενεκτικού συνεδρίου είναι απηχή μάλλον τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαχείριση του προϋπολογισμού, διότι η συνθήκη απαιτεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός να εκτελείται σε συμφωνία με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτείται ή καλείται να χορηγεί την απαλλαγή πάλι στην ε, βάση και των δύο αυτών στοιχείων, κανονικότητας και χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Για να γίνει αυτό δυνατό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει λογαριασμούς που θα δείχνουν πώς εισπράχθηκαν οι πόροι και πώς χρησιμοποιήθηκαν και από τότε που ισχύει η, συνθήκη της Λισαβόνας υποβάλλεται και έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ετήσιες και ειδικέ εκθέσεις ως συμπλήρωμα ενημέρωσης για το Κοινοβούλιο και επίσης εξασφάλιση της αξιοπιστίας. Το πώς ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του το Συμβούλιο είναι δική του ευθύνη. Το ίδιο το Συμβούλιο, το Συνέδριο συγγνώμη, ε, αποφασίζει όπως είπαν και οι ομολογοί μου προηγουμένως, ισχύει και εδώ η αρχή της θεσμικής ανεξαρτησίας. Και εδώ έχουμε τώρα στον δεύτερο λόγο για τον οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην διακρίνουμε υπερβολικά ανάμεσα στην απόδοση και στην αποτελεσματικότητα. Ο λόγος αυτός είναι ο επαγγελματικός. Το συνέδριο είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο όπως το GAO ή ο γαλλικός ε, αρμόδιος οργανισμός στην, εργαζόμαστε στην βάση διεθνών προτύπων που λέγονται ΙΣΑΙ και αυτά αποτελούν το σαφές πλαίσιο που είναι η βάση για την ερμηνεία που δίνει το συνέδριο στην εντολή του και για την άσκηση των καθηκόντων του. Αυτό το πλαίσιο των ΙΣΑΙ εντοπίζει τρία είδη ελέγχων. Οικονομικό, έλεγχο κανονικότητας και έλεγχο αποδοτικότητας. Θα τονίσω μονάχα και πολύ σύντομα περί πρόκειται. Ο οικονομικός έλεγχος καλύπτει την αξιοπιστία των εκθέσεων τη συμμόρφωσης ή κανονικότητας και της αποδοτικότητας εξετάζει την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της χρήσης των κονδυλίων οι ομολογοί μου μίλησαν για τις αρχές αυτές και πώς τις ερμηνεύουν αναπερίπτωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι ο έλεγχος συμμόρφωσης, νομιμότητας δηλαδή ή κανονικότητας μπορεί να εκτελεστεί και μόνος του ή και σε συνδυασμό με τους άλλους. Όποιος εξετάσει τις συνθήκες, δηλαδή τις ε, διατάξεις των συνθήκων, βλέπει ότι το, το συνέδριο συγγνώμη, επιλέγει την συνδυασμένη προσέγγιση οι δηλώσεις αξιοπιστίας του συνεδρίου είναι αποτέλεσμα ελέγχων ε, νομιμότητας που γίνονται στην βάση των, οικονομικών, των ελέγχων οικονομικών λογαριασμών. Περιλαμβάνουν κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις νομοθεσίας. Έτσι, από μια θεωρητική σκοπιά πρέπει να προσέχουμε να μην στοχεύσουμε υπερβολικά στις διαφορές ανάμεσα στα τρία είδη ελέγχων. Δεν είναι παρά εργαλεία που καλύτερα είναι να χρησιμοποιούνται όλα μαζί. Ο τρίτος λόγος για να μην δώσουμε υπερβολική έμφαση στις διαφορές αυτές είναι περισσότερο πρακτικού χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα θέματα ε, νομιμότητας και απόδοσης διασυνδέονται για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Οι έλεγχοι λοιπόν και οι εκθέσεις που υποβάλλουμε απηχούν το γεγονός αυτό. Για παράδειγμα, το συνέδριο με τους ελέγχους του δείχνει ότι σφάλματα στην κανονικότητα έρχονται σε περιπτώσεις όπου δεν επιτυχάνονται οι στόχοι ή που δεν γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, όταν πληρωμές κατευθύνονται σε μη επιλέξιμες δαπάνες. Και το ίδιο το συνέδριο χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων δηλώσεως αξιοπιστίας για να εντοπίσει τομείς όπου ίσως τίθεται σε κίνδυνο η αποδοτικότητα. Το συνέδριο επίσης διεξάγει ελέγχους αποδοτικότητας που οδηγούν σε παρατηρήσεις που περιλαμβάνουμε στις ειδικέ μας εκθέσεις όπου τονίζουμε θέματα που έχουν συνέπειες στην οικονομία, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Έτσι λοιπόν οι έλεγχοι αποδοτικότητας αποτελούν τη βάση για τις συστάσεις μας που περιλαμβάνουμε στις ειδικέ εκθέσεις ή σε γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών προτάσεων για το πώς να βελτιώσουμε δηλαδή το νομικό πλαίσιο για να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα. Και έτσι έρχομαι στον τελευταίο και πιο σημαντικό λόγο για να μην κάνουμε τις τόσο έντονα τις διακρίσεις αυτές, που είναι το δημόσιο συμφέρον. Δεν διεξάγουμε τους ελέγχους μας, ντάς ή άλλους, μόνο επειδή οφείλουμε. Τους διεξάγουμε επίσης διότι αυτοί συμβάλλουν στην αποτελεσματική λογοδοσία προς τον Ευρωπαίο πολίτη για κάθε ευρώ που εισπράτεται και δαπανάται μέσω του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Ο στρατηγικός μας στόχος για την περίοδο 2013 έως 2017 είναι να μεγιστοποιήσουμε την αξία της συμβολής του συνεδρίου στην βελτίωση της δημόσιας λογοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτεραιότητά μας είναι να στοχεύσουμε τα προϊόντα μας, το έργο μας, στην επίτευξη αυτού του στόχου. Από τη δική μας σκοπιά αυτό σημαίνει σύνταξη ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων που να βασίζονται στους ελέγχους μας και που να αντιμετωπίζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των ενδιαφέρομενων μερών μας, ιδίως του κοινοβουλίου σας και των πολιτών που εκπροσωπείτε. Ο Ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πού δαπανώνται τα χρήματά του. Δαπανώνται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκαν και δαπανώνται χρηστά, με χρηστό τρόπο. Αυτό σημαίνει ανάγκη αποτελεσματικών ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι, ότι γίνονται σεβαστοί οι κανόνες, οι δημοσιονομικοί κανόνες και ότι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, επιτυγχάνονται τόσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Όσον αφορά τους λογαριασμούς της Ένωσης, το συνέδριο τους έχει βρει αξιόπιστους για έναν αριθμό ετών τώρα. Το έργο του συνεδρίου που οδηγεί στις γλώσσες αξιοπιστίας έχει συμβάλει. Εμείς ταχθήκαμε υπέρ της χρήσης ενός σύγχρονου λογιστικού πλαισίου βασισμένου σε καταγραφές βάσει δημιουργίας υποχρέωσης ή αξίας και έχουμε κάνει σχετικές συστάσεις για την βελτίωση των λογιστικών συστημάτων και μάλιστα έχουμε επιτύχει. Όσον αφορά την κανονικότητα, εδώ η εικόνα είναι πιο περίπλοκη παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στους εσωτερικούς ελέγχους τα τελευταία χρόνια το συνέδριο συνεχίζει να διαπιστώνει, αγαπητοί βουλευτές, υψηλό σχετικά επίπεδο μη κανονικών πληρωμών. Το 2011 υπολογίζεται το ποσοστό σφαλμάτος σε 3,9%. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είναι αδύνατον να φτιάξει κανείς μια συνολική εικόνα. Οι δύο πρώτες εκδόσεις της έκθεσης αξιολόγησης κατέδειξαν ότι το, τα υλικά δεν έχουν μπει ακόμα στη σωστή θέση για να μπορέσει να αποτελέσει αυτό ένα σωστό εργαλείο για τον δημόσιο έλεγχο. Πολλά προγράμματα δαπανών εξακολουθούν ε, να στερούνται καθαρών στόχων και ε, σκοπών. Η δημόσια διαχείριση και ο έλεγχος προκύπτουν σήμερα από τις εξελίξεις που έχουν προέλθει από τις δυτικές μεταρρυθμίσεις της ε, Κομισιόν που έχει αρχίσει τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και περιλαμβάνει και αυτή ένα λογιστικό σύστημα βασισμένο στη, ε, στη δημιουργία αξίας με εσωτερικούς ελέγχους και μάλιστα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων και πάλι το έργο του συνεδρίου είτε η δηλώση αξιοπιστίας είτε ο έλεγχος αποδοτικότητας έχουν συμβάλει στην δημιουργία του πλαισίου αυτού. Η δική μας εμπειρία των ελέγχων αποτέλεσε τη βάση για την γνωμοδότησή μας για ένα πρότυπο ενίο ελέγχου στο οποίο περιλάβαμε τις ιδέες μας για το πώς πρέπει να είναι ένα τέτοιο πλαίσιο. Και έχουμε κάνει και τους σχετικούς ελέγχους τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχευε κυρίως στον έλεγχο της, της κανονικότητας των πληρωμών με στόχο να μειώσει το επίπεδο των μη κανονικών πληρωμών από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό σε κάτω του 2%. Όπως είναι το ίδιο ποσοστό και που το λέει ο κύριος Μιούλτερ τον μαγικό αριθμό. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, το συνέδριο έχει καταλήξει σε ένα υψηλό σχετικά ποσοστό σφάλματος. Από το 2006 αυτό το εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματος μειώνεται, γιατί το 2006 ήταν πάνω από 7%. Το 2011 ήταν 3,9%. Υπάρχουν βέβαια κάποιες διακυμάνσεις, αλλά αυτές εξηγούνται και από τεχνικούς λόγους. Όμως δεν θα επεκταθώ. Ίσως το Νοέμβριο να είναι καλύτερα. Όπως ξέρετε, το συνέδριο έχει τονίσει ότι από κάποια στιγμή και μετά το κόστος των ελέγχων αρχίζει και είναι μεγαλύτερο από το όφελος από την μείωση του ποσοστού σφάλματος. Γι' αυτό και ενθαρρύνουμε αυτούς που ασκούν την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό ορισμένων προγραμμάτων και από αυτή τη σκοπιά προβαίνει στην spending review, το προτείνει δηλαδή το συνέδριο που θεωρεί ότι πρέπει να είναι πιο στοχευμένη σε ο προγραμματισμός της Ένωσης. Το συνέδριο τονίζει ότι η στόχευση σε αποτελέσματα δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της κανονικότητας και γι' αυτό το λόγο αρχές του 2010 εκδώσαμε γνωμοδότηση ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην ποιότητα των δαπανών για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Κατά την άποψή μας, οι δαπάνες καλής ποιότητας σημαίνει ότι σέβονται τους κανόνες και επιτυγχάνουν αποτελέσματα. Νομιμότητα και αποδοτικότητα είναι δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αυτό είναι σημαντικό και έχει σημαντικές επιπτώσεις και για τον εσωτερικό έλεγχο, τον εξωτερικό έλεγχο, αλλά και για την πολιτική εποπτεία. Ιδίω αυτό το focus on results πρέπει να απηχείται σε τέσσερα σημεία. Οι ρόλοι της διαχείρισης και οι ευθύνε πρέπει να είναι ξεκάθαροι και απλοί. Στόχοι και σκοποί προς επίτευξη. Επίσης, καθαρή, σαφής και μετρήσιμη. Οι όροι πληρωμής για τους δικαιούχους. Και τέλος, οι απαιτήσει καταχώρησης, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων. Επίσης πρέπει να είναι ξεκάθαρα και απλά. Αυτά, εφόσον συμβούν, θα σημάνουν μια μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας των όσων λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις και των οικονομικών διαχειριστών και σημαίνει επίσης μεγάλη ευθύνη για ένα σχεδιασμό πιο αποδοτικών προγραμμάτων. Διότι την ευθύνη δεν φέρει μονάχα αυτός που κάνει τον τελικό έλεγχο. Πρέπει αυτοί που σχεδιάζουν τα συστήματα να γνωρίζουν τι ακριβώς επιθυμούν να επιτύχουν. Γι' αυτό και τώρα η νέα, προγραμμα... η προγραμματική περίοδος μας επιτρέπει να κάνουμε πρόοδο, βελτιώνοντας και την λογοδοσία για προγράμματα και σχέδια μετά το 2013 δίνοντας περισσότερη, περισσότερη στόχευση στα αποτελέσματα. Και αυτά νομίζω θα τα πει και ο κύριος Σέμετα. Με κύριες προτάσεις για τη Γεωργία, για παράδειγμα, έχω, που έχουμε υποβάλει συστάσεις εμείς και τις έχει, έχει, χρησιμοποιήσει το Κοινοβουλίο. Ως γνωρίζετε, κατά την άποψη του συνεδρίου, έχουν ήδη χαθεί κάποιες ευκαιρίες. Και μάλιστα στο υψηλότατο επίπεδο της ε, νομοθεσίας για να διευκρινιστούν ακόμα περισσότερο οι στόχοι, να απλοποιηθούν τα προγράμματα, να συνδεθούν οι πληρωμές με το αποτέλεσμα πιο στενά και να βελτιωθούν οι ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες για αλλαγή επί το θετικότερο και στα χαμηλότερα επίπεδα της νομοθεσίας και μάλιστα και όταν προγράμματα και σχέδια πρόκειται να εφαρμοστούν. Υπό το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, η χρηματοδότηση που δίνεται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό εξακολουθεί να είναι στην βάση, σε μέγα βαθμό, επιχορηγήσεων. Κατά την άποψη του συνεδρίου, θα πρέπει να, συνδεθεί, να συνδεθούν μάλλον τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την λήψη επιχορηγήσεων πιο στενά με το output, με τις εκροές, δηλαδή με τα αποτελέσματα. Άρα payment by results. Με το παράδειγμα που έδωσε ο κ. Σκυλακάκης, με εκείνο το λιμάνι που δεν έχει καράβια, θα πρέπει οι τελικές πληρωμές να συνδεθούν με την πραγματική έναρξη της χρήσης του λιμανιού. Αν τελικά συμβεί αυτό, η διαφορά μεταξύ κανονικότητας και αποδοτικότητας, δηλαδή νομιμότητας και αποδοτικότητας, θα είναι ακόμα πιο περιορισμένη από ό,τι τώρα. Έτσι, κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη, κατά την άποψή μας, το συνέδριο θεωρεί ότι ο έλεγχος δημοσιονομικός νομιμότητας και απόδοσης είναι ουσιώδη εργαλεία και βοηθούν εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πολιτική εποπτεία των οικονομικών της Ένωσης να απαιτούν λογοδοσία από τους υπεύθυνους διαχείρισης. Αυτό δε για το συνέδριο σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να διεξάγουμε ελέγχους και να συντάσσουμε εκθέσεις που βοηθούν το Κοινοβούλιο να ε, αντιμετωπίσει τις ευθύνες του. Και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο πάλι από τη μεριά του να κάνει την βέλτιστη δυνατή χρήση όλου του φάσματος των προϊόντων των εργασιών του συνεδρίου. Θα αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις ακόμη μπροστά μας. Για παράδειγμα, με την εισαγωγή νέων δημοσιονομικών εργαλείων. Εμεί μπορούμε να υποστηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έγγραφα θέσεων, με γενικέ επιθεωρήσει και με γνωμοδοτήσει που θα αναλύουν τι επιπτώσει των εξελίξεων αυτών για την ε, δημοσιονομική διαχείριση, για του ελέγχου και για τη λογοδοσία. Ωστόσο, του ελέγχου δεν του κάνουμε εν κενό. Θα μπορούμε να συνεχίσουμε να ασκούμε του ελέγχου στο μέλλον με το πώ και το τι θα εξαρτηθεί από το πώς θα αναπτυχθεί το πλαίσιο των εσωτερικών ελέγχων. Είναι σαφές ότι αυτό, το, αυτή η πυραμίδα αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει να ολοκληρωθεί. Πρέπει να δημιουργηθεί εκ των κάτω. Εάν η Κομισιόν είναι σε θέση να παράσχει επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες για το ποσοστό σφάλματος βασισμένη στις δηλώσεις αξιοπιστίας τα νούμερα αυτά μπορούν να σημάνουν σημαντική συμβολή για την DAS. Επίσης, οι στόχοι της αποδοτικότητας πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο διαχείρισης πριν να γίνουν κριτήρια του ελέγχου. Με τέτοιου είδους υλικά η αξιολόγηση, η έκθεση μάλλον αξιολόγησης της Κομισιόν του άρθρου 318 μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τον δημόσιο έλεγχο. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι το ολοκληρωμένο ιστορικό πλαίσιο ελέγχου προσφέρει και τις δυνατότητες για το συνέδριο να, να συνεργαστεί και με διεθνείς οργανισμούς ελέγχου. Αυτό μάλιστα είναι μια οδός την οποία σκοπεύουμε να εξετάσουμε προσεκτικά μαζί με, την, ε, με το Γαλλικό Ελεκτικό Συνέδριο αλλά και με τα, συνέδρια, τα συνέδρια των υπολείπων χωρών. Και η συνεργασία μεταξύ των υπά των οργάνων ελέγχου θα είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ευρωπαϊκή διαχείριση. Ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας και η δημοσιονομική και οικονομική επιτήρηση είναι δύο εργαλεία μέσα στο, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που θα επιτρέψουν και στο Κοινοβούλιο και στους πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα της αποδοτικότητας. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα αλλά πιστεύω ότι η βελτιωμένη λογοδοσία για την χρήση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και να σφυριλατηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνέδριο θα συνεχίσει να ασκεί τους ελέγχους του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την επίτευξη του στόχου αυτού. Θα σας προσφέρουμε αξιοπιστία και θα σας συνοδεύουμε σε κάθε σας ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ακούσαμε την άποψη λοιπόν του ελεγκτικού συνεδρίου και σημειώνουμε αυτά που είπατε για τον προσανατολισμό στον έλεγχο των επιδόσεων But let us η νομιμότητα των δαπανών από τη μία, αποτελεσματικότητα από την άλλη. Τώρα θα ακούσουμε και την άποψη του Επιτρέπου Σέμετα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Καλδέρα, κύριε και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Μου ζητήθηκε να μιλήσω με θέμα η χρήση των δικτών αποτελεσμάτων και η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές εδώ και κάποια χρόνια ο έλεγχος ε, αποτελεσμάτων έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Καλντέρα. Αυτό το καλωσορίζει η Κομισιόν καθώς τα αποτελέσματα αυτών έχουν μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για το τι κάνουν τα προγράμματά μας, ε, το πώς αποδίδουν καθώς βεβαίως και υποδείξεις για το πώς μπορούν να βελτιωθούν. Γι' αυτό χαρήκαμε για το ότι συζητήθηκε αυτό το θέμα και οι διάφορες πτυχές του. Ο λόγος σημασίας βεβαίως αυτών των ελέγχων είναι προφανής. Το νομικό πλαίσιο των ελέγχων προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στα αποτελέσματα αντί για τις ε, δαπάνες ε, και τα κονδύλια. Οπότε τα προγράμματα ελέγχου θα πρέπει να είναι σαφή και να αναφέρονται στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής. Επιπλέον, τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την περιοδική μέτρηση αυτών των αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις Κομισιόν για τη νέα προγραμματική περίοδο περιέχουν σαφή παραδείγματα αυτής προσέγγισης. Η οικονομική κρίση απαιτεί από όλους μας να υιοθετήσουμε μία προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών. Σε αυτούς τους δύσκολους ε, καιρούς, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 αποτελεί ένα σταθερό επενδυτικό ορίζοντα για να υπάρχει χρηματοδότηση για τους επενδυτές, για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Όμως οι όροι για επιτυχή προγράμματα είναι να εστιαστούμε στις σωστές προτεραιότητες και στα μέγιστα αποτελέσματα. Η Κομισιόν έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθυντήρες γραμμές για να διασφαλίσουμε πως η ποιότητα των δαπανών θα βελτιωθεί. Να αναφέρω δύο παραδείγματα. Πρώτον, οι στόχοι και το έβρος του προγράμματος ε, θα σχετίζονται άμεσα με τη στρατηγική 2020 για ανάπτυξη και δουλειέ. Όπω ανέφερα ήδη πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι προτεραιότητές μα με, γενικό, με τους γενικότερους πολιτικούς μας στόχους. Το πρασίνισμα τη γεωργίας είναι ένα παράδειγμα. Η θεματική εστίαση στα διαρθρωτικά ταμεία είναι άλλο. Δεύτερον, τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την μακροοικονομική πολιτική και τις προτεραιότητες που απορρέουν από αυτή. Πρέπει να διασφαλίσουμε πώς η πολύτιμη αυτή χρηματοδότηση θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ε, που αναφέρονται στις συστάσεις αναχώρα που κάνει η Κομισιόν και εγκρίνει το Συμβουλίο. Η Κομισιόν έχει σχεδιάσει τις ε, προτάσεις της για νέα προγράμματα στο Πουδεπού με στόχο να έχουμε ένα ισχυρότερο πλαίσιο απόδοσης. Οπότε έχουμε εστιαστεί στα αποτελέσματα και την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Γι' αυτό έχουμε τρία νέα σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, κάποιους βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με την κατάλληλη σύνδεση βεβαίως με τους στόχους του 2022. συμπεριλαμβάνει δείκτες που εστιάζουν στην προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την ε, αποτελεσματικότητα και το γενικότερο αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Τρίτον, το νέο πλαίσιο αυτό δημιουργεί ε, ένα πλαίσιο για αξιολόγηση για την παραγωγή των στον δεδομένων. Έτσι θα μπορούμε έγκαιρα να αξιολογούμε τα αποτελέσματα και την απόδοση και οι ελεγκτές θα μπορούν να ορίζουν καλύτερα τα κριτήρια ελέγχου με βάση τα οποία θα κρίνεται η απόδοση των μετρών. Ας δούμε τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία τα επενδυτικά για την περίοδο 2014-2020 ως παράδειγμα. Τι παρατηρούμε. Πρώτα απ' όλα ευθυγραμμίζονται τα προγράμματα δαπανών και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να στηρίζουν τη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Δεύτερον, ένα νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο που καλύπτει πέντε διαρθρωτικά ταμεία θα καθοριστεί για να υπάρχει μία συνέπεια μεταξύ των διαφόρων στόχων. Τρίτον, θα υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο απόδοσης έτσι ώστε για κάθε προτεραιότητα να υπάρχουν δείκτες και στόχοι ποιοτικοί και ποσοτικοί. Θα συμπεριλαμβάνουν οικονομικούς δείκτες ε, που θα αφορούν τις δαπάνες, δείκτες ε, αποτελεσμάτων και εκρών. Και τέλος, ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα βασίζεται σε αυτούς τους δείκτες ε, με συγκεκριμένες αξιολογήσεις εξ για το κάθε πρόγραμμα στην προγραμματική περίοδο και εξποστ post που θα εξετάζει την αποτελεσματικότητα και αποτελεσματική χρήση των ε, κονδυλίων. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στην κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήθελα τώρα να έρθω σε μια άλλη σχετική πτυχή η οποία είναι οι αναφορές. Το άρθρο 318 προβλέπει μια έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τη της Λισαβόνας. Από το οικονομικό έτος 2010 η Κομισιόν υποβάλλει συγκεκριμένες πληροφορίες απόδοση σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου του και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο η Κομισιόν εργάζεται συνεχώς για να βελτιώνει αυτές τις εκθέσεις. Το νέο πλαίσιο αυτό θα μας δώσει τα εργαλεία για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες ε, για πληροφορίες που ζητάει η αρχή απαλλαγής. Ο προσωρινός σχεδιασμός καθορίζεται σε ένα σχέδιο δράσης που είχε συμπεριληφθεί στην τελευταία έκθεση αξιολόγηση του έτους 2012. Προβλέπει πως οι πληροφορίες απόδοσης από τον κύκλο στρατηγικού σχεδιασμού της Κομισιόν θα εσωματώνται καλύτερα στην έκθεση αυτή. Όσο έχουν τα πράγματα, οι δείκτες ορόσημα και στόχοι που περιλαμβάνονται στα προγράμματα θα περιγραφούν στα διαχειριστικά σχέδια της Κομισιόν και μετά θα συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Τέλος, θα αξιολογηθεί η συνολική απόδοση στην ε, έκθεση αξιολόγησης. Έτσι θα διασφαλιστεί πως τα δεδομένα σε όλα τα προγράμματα δαπανών θα αξιολογηθούν με τρόπο ενιαίο. Αλλά έχουμε και άλλες βελτιώσεις κατά νου. Οι μελλοντικές εκθέσεις, παραδείγματος χάρη, θα έχουν ένα συνολικό πλαίσιο για παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων μέχρι το τέλος του επόμενου πι δελτα πι. Ένα πλαίσιο που αποτελείται από μια γενική έποψη των προγραμμάτων αυτών, τους βασικούς δείκτες ε, και την παρακολούθηση που θα γίνεται και βεβαίως τον χρόνο της αξιολόγησης. το πλαίσιο λοιπόν αυτής της έξυπνης αξιολόγησης η Κομισιόν θα εκδώσει νέες κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης για να ενισχυθεί η πολιτική αυτή αξιολόγησης και να ευθυγραμμιστεί με το νέο πλαίσιο απόδοσης. Κυρίε και κύριοι, όπως βλέπετε από αυτά τα οποία παρουσίασα, η Κομισιόν έχει ήδη αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να μετρήσει καλύτερα την απόδοση και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων μας. Ε, έχουν οριστεί δείκτες για το τρέχον πρόγραμμα και θα γίνει το ίδιο και για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Είμαστε προετοιμασμένοι να εφαρμόσουμε μια προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα και την απόδοση. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Commissioner. Now Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα ακούσουμε ερωτήσεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Πίπερ, ο οποίος ε, ζήτησε πρώτος τον λόγο. Έχετε τον λόγο. vielen Dank. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η παρέμβαση του Προέδρου του Συνεδρίου και του Επιτρόπου με εντυπωσίασαν με το βλέμμα σαφώς στραμμένο στο μέλλον σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διαφάνειας του ελέγχου της αποτελεσματικότητας χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν θα μπω στα όσα δεν συμφωνώ. Θα έρθω σε ένα θέμα όπου εγώ διαβλέπω μεγάλο κίνδυνο για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εάν όντω κάνουμε όσα εξήγησε μόλις ο Επιτροποσέμετα. Σέμετα. Μια χώρα μέλος ποτέ δεν θα τολμήσει να ελέγξει τα δημοσιονομικά κονδύλια με κριτήρια εάν μειώθηκε η ανεργία, εάν κάποιες επιχειρήσεις προέβησαν σε κάποια καινοτομία και μάλιστα να τολμήσει και να τα μετρήσει αυτά τα πράγματα. Τόσα έγιναν με τόσα λεφτά ε, στη βάση των τάδε δικτών. Αυτό για τη Γερμανία ή τη Γαλλία θα οδηγήσει σε καταστροφή. Γιατί αυτού του είδους οι πολιτικές υποσχέσεις είναι αδύνατο να τηρηθούν στις χώρες μέλη. Δεν θέλω να πω με αυτά τα λόγια ότι η προσέγγιση δηλαδή να αναπτυχθούν δείκτες για την απόδοση, την αποδοτικότητα είναι λάθος. Ε, να είναι δείκτες μετρήσιμοι, ασφαλώς η προσέγγιση αυτή είναι σωστή. Αλλά σας παρακαλώ, ας ρίξουμε το βάρος μας πραγματικά σε πράγματα που είναι όντως ευρωπαϊκής αρμοδιότητας, που όντως προσφέρουν μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Το παράδειγμα που αναφέρατε και εσείς, για παράδειγμα υποδομές, καινοτομίες σε επιχειρήσεις εφόσον αυτές προσφέρουν κάποια προστιθέμενη αξία. Αυτά όντως είναι μετρήσιμα. Αν πάρουμε τώρα τη λίστα των δικτών, κύριε Σέμετα, που έχει αναπτύξει ο συνάδελφός σας Άντορ, ορισμένες, ορισμένοι από τους αυτούς, αριθμός των αστέγων, ας πούμε, μειώθηκε ο αριθμός των αστέγων. Αν μειώθηκε τότε πετύχαμε πολλά με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Αριθμός των παιδιών κάτω των τριών ετών σε κέντρα παιδικής φροντίδας, σε ε, παιδικούς σταθμούς. Δείκτης που προτείνει ο κύριος Σάντορ. Εφόσον υπάρχουν περισσότερα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς κάτω των τριών ετών, αυτό σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί καλύτερα τα ευρωπαϊκά χρήματα. Εκεί έτσι θα μετράτε στο μέλλον η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός παιδιών με υψηλότερο απολυτήριο, δηλαδή ε, δίπλωμα που έχουν τελειώσει το σχολείο. Αν τελειώσουν αργότερα το σχολείο, στη Γερμανία για παράδειγμα, υποτίθεται ότι είναι επιτυχία, ευρωπαϊκή επιτυχία. Μα ε, κοιτάξτε, είναι δυνατόν ιδίω στην Νότια Ευρώπη διαπιστώνουμε προβλήματα ιδίω στα μέσα επίπεδα της εκπαίδευσης και όχι στην ανώτερη. Αυτά τα πράγματα που ανέφερα μόλις. Αριθμός των επισκεπτών θεατρικών παραστάσεων. Και αυτό είναι δείκτης, λέει. Αριθμός επισκεπτών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κοιτάξτε, προσοχή, κομισιόν και όλοι μας. Με τέτοιους δείκτες να πάμε να μετρήσουμε την ευρωπαϊκή επιτυχία κατά 98% αυτά τα πράγματα είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Είναι κλασική επικουρικότητα. Εκεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίπεδου κόκκου άμμου. Αυτά τα πράγματα όλα θα γίνουν, θα υλοποιηθούν και χωρίς ευρωπαϊκές πιστώσεις. Φοβούμε λοιπόν ότι ιδίω σε αυτούς τους κοινωνικούς τομείς, εγώ μάλιστα θα τα πω αυτά στην έκθεσή μου για την απαλλαγή της Κομισιόν, πλανάστε, πλανάστε εκτρά, διότι οδηγήστε σε μια κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία όπου θεωρούμε ότι μπορούμε βασισμένοι στις ευρωπαϊκές πιστώσεις να επιβάλλουμε στόχους και μετά από πέντε χρόνια να καθίσουμε να μετρήσουμε πόσα παιδάκια πηγαίνουν τώρα στους παιδικούς σταθμούς για να δούμε αν αποδίδουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εάν πάμε έτσι να μετρήσουμε την επιτυχία μας κυρίες και κύριοι, τότε θα αποτύχουμε παταγωδός. Γιατί με αυτά τα λίγα δις ευρώ που έχουμε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τον αποτελεσματικό τρόπο που θέλουμε. Και γι' αυτό θα πω και στον κύριο Καλντέιρα και στον κύριο Σέμετα. Σας παρακαλώ, λάβετε το υπόψη σας. Εμείς ζητήσαμε όντως δίκτες μέτρηση για την υποδομή. Αλλά τώρα να θέλουμε να μετρήσουμε την χρήση των ευρωπαϊκών πιστώσεων με βάση τέτοιου είδους κοινωνικούς δείκτες, εγώ το θεωρώ αυτό απόλυτα πεπλανημένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις πρώτα και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Ο κύριος Μπαλτσίτης έχει το λόγο. Μετά ο κύριος Κυλακάκης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεισφορά του στη σημερινή συζήτηση. Είναι σημαντικό βέβαια που ακούσαμε και τις εμπειρίες των άλλων κρατών. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνει κανείς ε, το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να, χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιηθεί το δημόσιο χρήμα. Πάντως είναι σαφές ότι βασικός μας στόχος είναι να γνωρίζει ο Ευρωπαίος πολίτης πόσο καλά χρησιμοποιούνται τα χρήματα που αυτός δίνει. Από την άλλη ακούσαμε ότι όταν χρησιμοποιούμε ε, πολλαπλούς δείκτες ε, στην ουσία ε, θα κινδυνεύουμε να γίνουμε μια προγραμματισμένη οικονομία όπως είπε κάποιος συνάδελφος. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη μέση οδό. Δεν θα πρέπει να παραμείνουμε σε απλά συνθήματα. Και φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι, κοιτάξτε, επειδή οι συνθήκες είναι δύσκολες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη σωστή χρήση του δημοσίου χρήματος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι τα κοινοτικά χρήματα δεν αρκούν για να λύσουν όλα τα προβλήματα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Λιθουανία έχουμε πολλαπλά θέματα και ε, τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά σε ορισμένους τομείς τους οποίους έχουμε προβλήματα είναι πολύ λίγα για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να τα ξεπεράσουμε. Οι στόχοι λοιπόν τους οποίους πρέπει να έχουμε ίσως θα πρέπει να είναι λιγότεροι γιατί τότε θα είναι πιο εύκολος ο έλεγχος των χρημάτων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Ξεκάθαροι στόγοι, μετρήσιμοι στόγοι και επίσης ε, με, ε, μετρήσιμες μέθοδοι για να υπολογίσουμε το κατά πόσον τους έχουμε πετύχει. Αυτό θα διασφαλίσει την αποδοτικότητα των προσπαθειών των ελεγκτικών συνεδρίων που έτσι και αλλιώ κάνουν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Έχουν δαπανηθεί πολύ, πολλά χρήματα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αιτήσια βάση Κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν σωστά, κάποια λιγότερο σωστά και θα χρειαστούν φυσικά πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία έχουμε. Δεν νομίζω ότι θα σταθούμε ποτέ ικανοί να μετρήσουμε τα πάντα με ακρίβεια. Θα πρέπει όμως να γίνουν ορισμένες προτάσεις και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε κάποια πράγματα να αλλάξουν σε σχέση με τον καθορισμό των στόχων, είτε των κοινωνικών στόχων, είτε των στόχων στον τομέα της ενέργειας, είτε των στόχων στον τομέα των μεταφορών. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει ε, να κρίνουν αν οι στόχοι αυτοί θα ε, ε, μπορέσουν να μετρηθούν με σωστό τρόπο και να εγγυηθούν έτσι τη σωστή χρήση των ποσών που είχαν διατεθεί. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσει ήδη σε μια πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει σωστά τους στόχους και πριν ορίσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να εξετάσει αν μπορεί πράγματι να ελέγξει σωστά τη διαδικασία επίτευξης των στόχων αυτών. δεν μπορούμε εμείς να προσπαθούμε να ελέγξουμε κάποιες διαδικασίες και από την άλλη βέβαια και εδώ είναι ένα άλλο θέμα τα κράτη-μέλη να μην μας δίνουν τα στοιχεία τα οποία είναι προαπαιτούμενο για να το πετύχουμε. Αυτό είναι σαν να έχουμε πέσει σε έναν μονόλογο ε, και μέσα από τον μονόλογο δεν θα μάθουμε τίποτα βέβαια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σκυλακάκης έχει το λόγο. Thank you and... Uh, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον, πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία ερώτηση καταρχάς προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορά με τους τομείς υψηλού κινδύνου. Είδαμε, ακούσαμε πως στις Ηνωμένε Πολιτείες εφαρμόζεται μια στρατηγική ε, για τον σωστό εντοπισμό των ε, τομέων υψηλού κινδύνου ε, όπου απαιτείται να αναλυθεί περαιτέρω δράσης από άλλες ίσως υπηρεσίες και στην περίπτωσή μας από την Επιτροπή ή το Συνέδριο. Έχετε λοιπόν υπόψη σας ότι αυτή η πρακτική ανείχνευσης και εντοπισμού των επικίνδυνων τομέων πρέπει να προωθηθεί γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ τον τρόπο με τον οποίο ασχολούμεθα με τα πράγματα. Μία δεύτερη παρατήρηση τώρα έχει σχέση με το εάν ο τρόπος με τον οποίο προσμετράμε τα πάντα θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικός. Βέβαια, αν συμπεριλάβουμε στους στόχους μας πράγματα που δεν μπορούμε να πετύχουμε, τότε προφανώς δεν θα πετύχουμε, είναι σαφές. Αλλά ήδη έχουμε αποτύχει. Ξέρουμε ότι το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρώπη, ανεργίας να το πω καλύτερα, είναι μια καταστροφή και μάλιστα σε ορισμένες χώρες μια τρομερή καταστροφή. Αλλά στροφοκαμιλίζοντας και ε, κρυβόμενοι ε, πίσω από την εθνική κυριαρχία είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα προσφέρει και σίγουρα δεν θέλουμε να φύξουμε την εθνική κυριαρχία, δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Κανένας δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική κυριαρχία και επικαλούμενος, επικαλούμενος την κυριαρχία αυτή την εθνική να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδιαίτερα σε ένα δημοσιονομικό περιβάλλον όπως είναι αυτό το σημερινό. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πιθανή σύγκρουση ανάμεσα στην εθνική κυριαρχία από τη μία και την δημοσιονομική ε, ολοκλήρωση από την άλλη το δημοσιονομικό περιβάλλον από την άλλη, ιδιαίτερα όταν, ε, τα, όταν τα, ομοσπονδιακά χρήματα, δηλαδή στην περίπτωση μας τα κοινοτικά χρήματα, είναι αυτά τα οποία θα καταστήσουν πιο καλή και πιο λειτουργική αυτήν την δημοσιονομική Ευρώπη. Και αυτό γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Και τώρα λέμε εμείς ότι ίσως δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να το υπολογίσουμε αυτό. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στο μέλλον. Αν δεν τολμήσουμε καν να προσμετρήσουμε αυτή, την, αυτό το στοιχείο, πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Να σας θυμίσω τις προσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχαμε πει ότι θα γινόμασταν η πιο ανταγωνιστική και η πιο καινοτόμα οικονομία στον κόσμο. Ε, δεν ε, ορίσαμε τρόπους υπολογισμού ε, της προσπάθειας επίτευξης των στόχων αυτών και φυσικά και αποτύχαμε. Thank you very much for comments, Jean-Pierre Ευχαριστώ Ζαν Πιέρο Ντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καθώς επίσης ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους, τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Μπερτράν και τον κύριο Μιμ για τις παρεμβάσεις σας. Ως Ευρωβουλευτής και επικειμένων των ευρωεκλογών έχω μια ανησυχία. Διερωτώ με εάν με όλους τους εκλεγμένους άρχοντες, ε, κυβερνήσεις, ε, το, τους δημόσιους λειτουργούς. Έχουμε άραγε προβληματιστεί αρκετά για την ε, αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των δημοσίων δαπανών. Εδώ μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια εγκύπτουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς. καθώς επίσης και, ε, ε, και τμήματα των περιφερειακών. Τώρα, στο επίπεδο εθνικό, ε, ευρωπαϊκό και περιφερειακό δεν έχουμε συνολική εικόνα. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι οι πολίτες έχουν λίγο το αίσθημα ότι καθίστανται μάρτυρες μιας σπατάλης ανεξέλεκτων δαπανών. Εγώ έχω κάνει παλαιόθεν μια πρόταση αλλά σας την υποβάλλω ξανά. Δεν θα ήταν δυνατό τώρα που γίνονται σπάνιοι οι δημόσιοι πόροι να προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν έλεγχο σχετικά με τις οικονομίες, με τις οικονομίες που μπορούμε να κάνουμε εάν τα βάλουμε, τα κάνουμε αμοιβαία, χωρίς να αγγίξουμε την ε, κυριαρχία των χωρών μελών, γιατί κάτι τέτοιο είναι αδυνατόν τώρα, αλλά ε, συνδυάζοντας τις δαπάνες. Εγώ ε, ασχολήθηκα με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και την ε, ενδιάμεση αναθεώρησή του. Μας είπαν ότι 15 φορές χρηματοδοτούνται ορισμένα έργα στις χώρες μέλη χωρίς κανένα συντονισμό. Διπλωματία. Έχουμε εκατοντάδες ακίνητα σε όλο τον πλανήτη με τις, ε, εκπροσω... με τις αντιπροσωπείες της Κομισιόν, τις ε, μας που δεν μοιράζονται ούτε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. Επίσης τώρα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν το θέμα της άμυνας. Ελπίζω να το συζητήσουν το θέμα αυτό, διότι είναι ε, οι, ε, οι ε, προπολογισμοί της άμυνας εντάσσονται στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Κάποια στιγμή δεν θα έχουμε δυνάμεις να μπορέσουν να υπεραμεινθούν της ευρωπαϊκής επικράτειας. Επίσης, οι εξωτερικές σχέσεις, ανάπτυξη, οι χώρες μέλη δίνουν αναπτυξιακή βοήθεια, η Ένωση επίσης. Δεν νομίζετε ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ένα είδος ελέγχου του συνδυασμού των εξοικονομήσεων που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να αγγίξουμε την ε, κυριαρχία των χωρών μελών, να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών στα τρία επίπεδα. Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτος μέλος, περιφέρεια και επομένως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εθνικές κυβερνήσεις και περιφερειακές εκτελεστικές αρχές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συνεργασία με τα Εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια να γίνει η έκθεση αυτή να υποβληθεί σε όλες τις γλώσσες εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συζητηθεί μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού για να εγγύψουμε και να απαντήσουμε στο ερώτημα Έχουμε αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των έργων, αλλά για όλες τις δημόσιες δαπάνες, όχι μόνο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όχι μόνο της ε, τάδε περιφέρειας ή της ε, τάδε κυβέρνησης, αλλά του συνόλου των δημοσίων δαπάνων, διότι όπως είπα τώρα που υπάρχει τέτοια σπάνιδα δημόσιων πόρων, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να φτάσουμε να συνεργαστούμε έχω την εντύπωση ότι εξακολουθώ είμαι εντός θέματος, γιατί το θέμα είναι η έλεγχη της νομιμότητας και της αποδοτικότητας των δαπανών. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ ωστόσο βλέποντας απέναντί μου αυτές τις υψηλές προσκεκλημένες προσωπικότητες να εκφράσω τα αισθήματα που με διέπουν ως αντιπρόσωπο των πολιτών και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Thank you very much, Jean-Pierre Audi. I see Σε ευχαριστώ, δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει τον λόγο οπότε να σας υπενθυμίσω πως έχουμε ακόμα α, παραπάνω από μισή ώρα στην διάθεσή μας λοιπόν κύριε Καλδέρα κύριε Επίτροπε θα ήθελα να σας ρωτήσω να σας ζητήσω ξανά να μας πείτε την απόψή σας, να πατήσετε στις ερωτήσεις, ε, σε αυτά τα οποία είπε ο Ζανπιέρη, ο κ. Μπαλτσίτης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τα σχόλια που έγιναν. Θεωρώ πως η παρατήρηση του κυρίου Πίπερ αφορούσε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θυμάται την αρχή της επικουρικότητας και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί επί του προϋπολογισμού της, του δημοσιονομικού πλαισίου, επί πολιτικών υπάρχει μία αρχή ε, που λέγεται προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, δεν είναι δουλειά των ελεγκτών να πούνε ποιες είναι οι προτεραιότητες οι πολιτικές ή τα μέσα ή οι δείκτες που θα μετρήσουν εμείς μπορούμε να κάνουμε τον ελεγχό μας ε, επί των αποτελεσμάτων ε, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν οριστεί και άρα η αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων πρέπει να μετριέται με βάση αυτά τα οποία συμφωνούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και τα σχετικά μέσα βέβαια. Αυτό το οποίο είπε ο κ. λέτε πως ε, χρειαζόμαστε κάτι το οποίο θα μας δίνει μια γενική εικόνα για, τη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, πράγματι σε κάποιους τομείς και αν δούμε τη διαρθρωτικά ταμεία, την πολιτική συνοχή. Ε, ναι, η συγχρηματοδότηση είναι σημείο κλειδί. Υπάρχει εθνικός προπολογισμό, αλλά υπάρχει και ευρωπαϊκός. Και πράγματι υπάρχει ένας ε, συμφωνημένος στόχος, ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και η Κομισιόν προτείνει νομίζω ένα μέσο, ένα εργαλείο, γιατί οι δείκτες αυτή η απόδοση δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι μέσα εργαλεία που ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να τα χρησιμοποιούν βεβαίως οι διαχειριστές για να παρακολουθούν, να προσαρμόζουν, να αλλάξουν ε, κάτι αν χρειάζεται και μετά βεβαίως οι ελεγκτές λένε ναι χρησιμοποιήστε αυτό αλλά ίσως χρησιμοποιείτε λάθος πράγμα. Ξεχάσατε το χύψη και όταν είχατε σχεδιάσει την πολιτική κάτι δεν είχε καλυφθεί από τους δείκτες οπότε υπάρχει ένα κενό. Εάν λοιπόν το δούμε ως μέσον για την καλύτερη χρήση των ε, κοντιλίων αυτών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλό των ε, δικαιούχων νομίζω μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τρόπο βέλτιστο σεβόμενοι βεβαίως πάντα τη, τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης τι είναι αυτό το οποίο καλύτερα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη δηλαδή την επικουρικότητα και βεβαίω οι στόχοι και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 πράγματι εκεί πέρα δημιουργεί κάποια πολυπλοκότητα. Δηλαδή ορίζονται στόχοι ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο με κάποια χρηματοδότηση που δεν είναι οπωσδήποτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά ζητάμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν εθνικά προγράμματα που χρηματοδοτούν κιόλα. Οπότε αντιλαμβάνουμε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Πίπερ αλλά προσπαθούμε επιτύχουμε κάτι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πω εγώ τώρα αν είναι σωστή η ε, στόχη της πολιτικής. Αυτό είναι θέμα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Απλά να θέσουμε τα πράγματα εντός σωστού πλαισίου. Τι μπορεί να κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Να δούμε. Είναι σωστή, ε, με συγχωρείτε, σαφής, ε, ξεκάθαρη η στόχη. Οι διαχειριστές ε, έχουν αντιδράσει ε, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έχουν προσαρμόσει τους ε, στόχους που είχαν αρχικά τεθεί. Ο κύριος Σκυλακάκης έθεσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Τι γίνεται... Ναι την ε, Ιρλανδία. Το 2010 είχαμε βγάλει ένα σχετικό έγγραφο, ε, πέρασε απαρατήρητο. Στο έγγραφο αυτό επιστήσαμε την προσοχή του Κοινοβουλίου και της Βουλικής Κομισιόν στα απλά αυτά ζητήματα που ανέφερα και που ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή, πρέπει τα προγράμματα να είναι απλά, μην περιπλέκουμε τη ζωή μας. Γιατί είναι και υψηλού κινδύνου κάτι τέτοιο. Και αυτός ο οποίος ε, μπορεί να το αλλάξει είναι αυτοί οι οποίοι συντάσσουν την ομοθεσία. Οπότε, είπαμε, να είστε προσεκτικοί, μην κάνετε τα πράγματα πολύ περίπλοκα, γιατί αν τα κάνετε πολύ περίπλοκα υπάρχει υψηλός κίνδυνος για ε, παράτυπες πληρωμές, ε, για ε, να είναι περίπλοκα τα αισθήματα εσωτερικού ελέγχου. Δεύτερον, σαφείς ευθύνες και κανόνες εφόσον υπάρχει επίπεδο ε, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό, τοπικό. Οπότε πρέπει να είναι σαφές το ποιος κάνει τι και ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Εάν δεν είναι σαφής η στόχη και κατανοητή από όλους, Βεβαίω τότε υπάρχει κίνδυνος. Θα έλεγα πως δεν ξεχνάμε πως ε, όταν υποβάλλουμε αυτή την πρόταση είχαμε αλλαγή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλάμβανε και ανέλαβε και ένα νέο κοινοβούλιο οπότε θεωρούσαν πως με την ευκαιρία ενός ε, νέου κοινοβουλίου, νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν καλή στιγμή να ευστήσουμε την ε, προσοχή σε αυτό το οποίο θεωρούσαμε κίνδυνο ε, για το γενικότερο πλαίσιο. Και αυτή τη στιγμή βεβαίω εξετάζουμε τη γενικότερη κατάσταση. Οπότε θα έλεγα πως ε, είμαστε μπροστά σε μια νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 ε, του χρόνου έχουμε και ευρωεκλογές νέος επίτροπος, νέα κομισιόν οπότε είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε το ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε πως έτσι αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες σας και βεβαίως αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και μπρο. Ε, είμαστε στη διάθεσή σα. Με συγχωρείτε να μακρηγόρησα. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος ότι είναι σωστά, πράγματι, ακόμα και σήμερα η Επιτροπή συζήτησε μια έκθεση για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. και θεωρούν πως η συνεργασία με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια ε, σε όλους τους τομείς είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Και ε, τόσο απλό είναι. Ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο υπονοεί οικονομικό συντονισμό, ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν υπόψη τι συστάσει του Συμβουλίου και τη Κομισιόν. Η Κομισιόν πρέπει να το παρακολουθεί αυτό, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα. Χρειαζόμαστε και τα υπόλοιπα ελεγκτικά συνέδρια και αυτό που θα να κάνουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, μην ζητάτε συγγνώμη. Μόνο θετικά βεβαίω μπορεί να είναι τα όσα μας είπατε και εξάλλου ήταν και πολύ ενδιαφέροντα. Κύριε Σεμέτα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να απαντήσω στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ, τον κύριο Σκυλακάκη και τον κύριο Μπαλτσίτης και για τα θέματα που έθεσαν σε σχέση με τους δείκτες. Εγώ ίσως και αντίθετα από τον κύριο Καλτέρα δεν βλέπω να υπάρχει μια αντίφαση στις παρατηρήσεις αυτές. Πρώτον, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αντίθετα με άλλες νομικές δικαιοδοσίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια περιφερειακή δομή η οποία βασίζει τον προγραμματισμό της σε νομοθετικές ρυθμίσεις και στην παρούσα φάση διαπραγματεύεστε πολλαπλές νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα της συνοχής, της κοινή αγροτικής πολιτικής όπου ήδη έχουμε καταλήξει σε ένα συμβιβασμό και γενικά βασίζουμε τις δαπάνες μας ε, σε νομικές αποφάσεις, σε νομικές πράξεις. Και για το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχει μια θα έλεγα πιο ολοκληρωμένη διαδικασία καθορισμού των στόχων στην οποία όλοι οι νομοθέτες ε, ε, συμφωνούν και περιλαμβάνονται επίσης και οι λεγόμενοι κομβικοί δείκτες και θα πρέπει οι συνομοθέτες να διαπραγματευθούν εάν πράγματι, να πούν εάν πράγματι συμφωνούν με τις προτάσεις τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν θέλουν να κρατήσουν τους δείκτες επιδόσεων. Ε, με βάση τους οποίους ε, το ελεγκτικό συνέδριο θα κάνει τους υπολογισμούς του, θα κάνει τους λογαριασμούς του και θα βλέπει αν θα είναι αποτελεσματικός ο τόπος αυτός. Πάντως θα πρέπει και για μια ενδιάμεση περίοδο να ισχύσουν οι δείκτες αυτοί έτσι ώστε να μην καταλήξουμε στο τέλος της δημοσιονομικής περίοδου συνειδητοποιώντα ότι λεγόμενοι κομβικοί, κομβικοί δείκτες στον τομέα της συνοχής σαν παράδειγμα είναι ανέφικτοι και τα χρήματα έχουν ήδη πλέον δαπανηθεί και δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται να δημιουργηθεί και μια πυραμίδα ενδιάμεσων δείκτων που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους τελικούς δείκτες ε, στους οποίους θα έχουν συμφωνήσει οι συνομοθέτες. Συμφωνώ με τον κύριο Πίπα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, παρεμβατικοί σε τομείς όπως οι δείκτες, οι λεγόμενοι αναπτυξιακοί κτλ. Και πράγματι υπάρχει η λογική που λέει ότι θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των δικτών που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενιοποιήσουμε την διαδικασία αυτή με στόχο την επίτευξη των αποτελεσμάτων που έχουμε στο τέλος των κεντρικών κομβικών λεγόμενων δικτών. Υπάρχουν δείκτες οποίους αναφερθήκατε σχετικά με την κοινωνική πολιτική. Φυσικά έχουμε και το κοινωνικό ταμείο στον τομέα αυτό, το οποίο θα πρέπει να δαπανά τα διαθέσιμα κονδύλια επί τη βάση των στόχων στους οποίους έχουν συμφωνήσει οι συνομοθέτες και επί τη βάση συγκεκριμένων δικτών. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι επιμέρους πιο συγκεκριμένοι δείκτες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί για το εάν πράγματι θα πρέπει να υιοθετήσουμε και επιπλέον δείκτες οι οποίοι θα είναι ειδικοί για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και βέβαια εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με τα ευρωπαϊκά χρήματα για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Τα χρήματα τα ευρωπαϊκά είναι περιορισμένα και τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν πολύ περισσότερα χρήματα για κοινωνικούς στόχους. Οι δείκτες λοιπόν και στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να είναι σχετικοί και με τα σύνολα ποσά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας προς ε, ε, τους συγκεκριμένους στόχους και σε σχέση με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Στον κοινωνικό τομέα πάντως το κοινοτικό χρήμα λειτουργεί ε, διευκολυντικά των ενεργειών στο εσωτερικό των κρατών μελών γιατί το σύνολο των ποσών που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περιορισμένο. να απαντήσω εδώ και στον κύριο Μπαλτσίτης. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε όλα τα επίπεδα του κύκλου στρατηγικού προγραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να πετύχουμε τους στόχους και να χρησιμοποιήσουμε τους κομβικούς δείκτες μέσω του καθορισμού εθνικών στόχων και ε, ετήσιας χρήσης δείκτων και μετά ε, τα αποτελέσματα αυτά να συμπεριληφθούν και να αντικατοπτρίζονται σωστά στις, ετήσιες, στις εκθέσεις αιτήσια δραστηριότητάς μας. και οι συνολικές εκθέσεις θα βασίζονται σε όλες αυτές τις αλήσους δικτών και οι εκθέσεις αξιολόγησης έτσι λοιπόν με τέτοιο τρόπο θα έχουν μεγαλύτερη και υψηλότερη γενικά ποιότητα. Ξεκινήσαμε γύρω στο 2010 με τις εκθέσεις αυτές, θέλουμε περισσότερο χρόνο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, εργαζόμαστε σκληρά και ήδη νομίζω έχουμε πετύχει μια ε, ε, ένα υψηλό επίπεδο και μπορούμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Έρχομαι σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Οντί τώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, πιθανές ε, επικαλύψεις σε περιπτώσεις συγκεκριμένων μείων των ε, δαπανών. Οι κανόνες μας απαγορεύουν τις επικαλύψεις αυτές και όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με μη αποδοτικές δαπάνες. Το 7ο πρόγραμμα σαν παράδειγμα μπορεί να σημειωθούν κάποιες επαναλήψεις δαπανών και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χαρακτηριστούν σαν μη αποδοτική μορφή δαπάνης. Σε κάποιους άλλους τομείς όπως η διπλωματική υπηρεσία, η, η άμυνα, είπατε και εσείς και συμφωνώ και εγώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα της άμυνας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει πολλαπλές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό και θα συζητηθούν στο Συμβούλιο σύντομα, το Δεκέμβριο. Πάντως εδώ τίθεται και ένα θέμα πολιτικό και μπορούμε εμείς να κάνουμε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και να παρουσιάσουμε τα καλύτερα δυνατά τεκμήρια για το καλό των ευρωπαϊκών πολιτικών σε συγκεκριμένους τομείς όπως η διπλωματική υπηρεσία και όπως η άμυνα. Αλλά είναι πολιτικό το θέμα, το θέμα τίθεται εδώ πράγματι της εθνικής κυριαρχίας και αν τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα ε, στην παρούσα φάση να προχωρήσουν. Ακριβώς στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη όρεξη από τα κράτη-μέλη να εκχωρήσουν περαιτέρω κυριαρχία στους τομείς αυτούς. Αλλά σιγά σιγά είδαμε ότι στον τομέα της άμυνας μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν αυτά κύριε Πρόεδρε, απάντησα στις ερωτήσεις σας νομίζω. Thank you very much. Ο Προεδρεύων, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι τα σχόλιά σας ήταν επαρκέστατα και επιστικά. Έχω τώρα το καθήκον να ερωτήσω τον αξιότιμο κύριο εισηγητή. Αν εσείς κύριε Σκυλακάκη επιθυμείτε να σχολιάσετε, μας μείνουν λίγα λεπτά. Νομίζω μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ακρόαση, απαντά ο κύριος Σκυλακάκης, που ε, είπα και πριν ότι είναι πολύ χρήσιμη. Ας ολοκληρώσω λέγοντας ότι διδαχθήκαμε πρώτα για το τι κάνουν άλλοι όπως οι Ενωμένε Πολιτείε, το γεγονός ότι αρχίζουμε τώρα αυτή την προσπάθεια που είναι βασισμένη στην αποδοτικότητα ενώ στις Ενωμένε Πολιτείες αυτό γίνεται εδώ και καιρό αυτό έχει και σχέση με τα ποσά των κονδυλίων που δαπανούμε και που είναι λιγότερο από 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω μιλείται για περίπου το 15 πλάσιο. Είναι προφανές λοιπόν ότι όντως οι Αμερικανοί είναι πολύ πιο προχωρημένοι ε, σε ό,τι αφορά την εξέταση των δαπανών στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να εξετάσουμε. Θα επανέλθω στους τομείς υψηλού κινδύνου, διότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα είπε ο αγαπητός πρόεδρος Καλντέρα. Εγώ μιλώ για συγκεκριμένους τομείς δαπανών γεωγραφικά χαρακτηρισμένους, όπου ίσως υπάρχουν αυξημένα προβλήματα. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να πείσει κανείς τους Ευρωπαίους πολίτες να δαπανίσουν περισσότερα χρήματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι διέπονται από επιφυλάξεις για το πώς δαπανώνται τα χρήματα αυτά και κυρίως οι χώρες οι οποίες είναι καθαροί εισφορείς. Ταυτόχρονα, άλλες χώρες που συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια και είναι λιγότερο στραμμένες στις εξαγωγές, ας το πω έτσι. Άρα δεν εποφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά. Και αυτές έχουν συμφέρον να δαπανηθούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Διότι το χρήμα θα λείψει τα επόμενα 7 χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για κοινή προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη. θα πρέπει να αρχίσουμε από μια μέτρηση των πραγμάτων. Κανένας δεν μπορεί να πει πώς έχει δαπανίσει τα πράγματα αν δεν έχει ξεκινήσει από μια μέτρηση του τι έχει κάνει. Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η πρώτη βάση για τους δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας. Πρέπει να μετρήσουμε λοιπόν. Ο κύριος Πίπερ βέβαια έχει αποχωρήσει από την αίθουσα, αλλά εξέφρασε τι επιφυλάξει του. Πρέπει να μετρήσουμε πράγματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις δαπάνες που έχουμε κάνει. Να μην πάμε να μετρήσουμε πράγματα που είναι σχεδόν αδύνατο να εξεύρει κανείς την διασύνδεση μεταξύ των δαπανών και της απόδοσης. Διότι αν πάτε να το κάνετε αυτό, μπαίνετε σε ένα χώρο όπου δεν έχει νόημα η μέτρηση. Να μην βάλουμε λοιπόν στα πρότυπα απόδοσης και για τους λόγους που εξήγησε ο κ. Πίπερα, αλλά και για λόγους τακτικής. Να μην βάλουμε λοιπόν πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Όμως μπορούν ακόμα πολλά πράγματα να μετρηθούν. Αν κάνουμε όμως ακριβώς αυτό. Δηλαδή πούμε μπορούμε ας πούμε να μετρήσουμε και τις εθνικές αποδόσεις. Βέβαια θα είναι κάτι όπου θα δοκιμάζουμε και ενδεχομένω να ασφάλουμε και να ξαναδοκιμάσουμε. Νομίζω ότι το συνέδριο μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη βοήθεια στην προσπάθεια αυτή. Πρέπει να καταστήσουμε όσο γίνεται πιο γνωστές τις ειδικές εκθέσεις και ελπίζω και ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αλλά και ως Κοινοβούλιο ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την δουλειά που κάνετε για να βελτιώσουμε τον τρόπο που ξοδεύουμε τα χρήματα άλλων. Μου φάνηκαν θετικά τα σχόλιά σας κύριε Σιγητά. Να πω τώρα ότι αισθάνομαι να είμαι μεταξύ βετεράνων της Επιτροπής όπως ο Ζανπιέρ, ο Γιάννη. Για μένα είναι η δέκατη διαδοχική χρονιά φέτος στην Επιτροπή αυτή. Και για πρώτη φορά ακούω μήνυμα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να, που να λέει ότι όλα θα πρέπει να είναι performance oriented. για να επιτευχθούν οι στόχοι να είναι αποδοτικοί και ταυτόχρονα να ικανοποιούν τα σχετικά πρότυπα. Αυτό δεν είναι λόγια βέβαια μόνο, αλλά απαιτεί και μια ανταπόκριση από την Κομισιόν. Και αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Σέμετα σήμερα είναι διαφορετικά από αυτά που ακούμε συνήθως από τους επιτρόπους. Δηλαδή μια επιτροπή η οποία προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στο ελληνικό συνέδριο. Ακούσαμε σήμερα πράγματα από δύο σημαντικούς ανεξάρτητους θεσμούς που όμως κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Η ακριβή έλεγχη είναι η απόδειξη του ύψου του επίπεδου εμπιστοσύνη, είπε κάποιο κάποτε. Όλα θα πρέπει να ελέγχονται και η τελευταία δεκάρα και το τελευταίο λεπτό του ευρώ προέρχεται από το δημόσιο, από την Ευρώπη δηλαδή, θα πρέπει να ελέγχεται. και σε ανταπόκριση σε κάθε πληροφορία, πληροφορία όποια από πού και αν προέρχεται αυτή. Αυτά είναι λογικά. Όμως ρωτώ, πώς θα βάλουμε ελεγκτές να ελέγχουν τους ελεγκτές. Όχι, Σας ευχαριστώ πάντως όλες και όλους για μια πραγματικά χρήσιμη και εντυπωσιακή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Καλντέρα, ευχαριστώ κύριε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε Καλντέρα, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε ε, Σέμετα, καθώς επίσης και τους κύριους Μπερνάρ και Μιμ για την τεχνογνωσία σας, για τις εμπειρίες σας, για τις απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστώ φίλοι Ευρωβουλευτέ που μείνατε μέχρι τέλους της αγοράσεως. διακόπτει τη συνεδρίαση. Thank you for